Ladies and gentlemen, please be seated. We start. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε και καλησπέρα σας. Δεύτερη εβδομάδα συνεδρίας της Υποεπιτροπής. Έχουμε τρεις, τρία θέματα εξαιρετικά σημαντικά στην ημερήσια διάταξη. Ξεκινώντας λοιπόν θα ήθελα να εγκριθεί η ημερήσια διάταξη για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται και όσοι ήθιστε σας ενημερώνω ότι έχουμε μετάδοση από το διαδίκτυο. Προτεραιότητα για τη διερμηνία δίνεται στις γλώσσες των μονίμων των τακτικών μελών της Υποεπιτροπής. Το επισημαίνω. Καθώς είχαμε κάποια προβλήματα σε σχέση με τη Σλοβακική, αλλά λύθηκε από ό,τι ξέρω. Υπάρχει η δυνατότητα για τη Σλοβακική. Εγκρίνουμε αν έχετε την καλοσύνη τα πρακτικά της υποεπιτροπής μας στις 16 Μαρτίου. Εάν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Και προχωρώ τώρα στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Με χαρά καλωσορίζω τον εκπρόσωπο της ε, αποστολής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σομαλία, τον, τον ταξιέρχο Αντώνιο Μάτζη. Η σημερινή μέρα όμως είναι γεμάτη. Θλίψη λόγω της δεύτερης μεγάλης μαζικής δολοφονίας στη Σομαλία. εργαζομένων από τις υπηρεσίες των ΗΕ που εκτελέστηκαν, που έχασαν τη ζωή τους και ίσως να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις. Είχαμε ακόμη την προηγούμενη εβδομάδα φόνους κοντά σε κτίρια της κυβέρνησης και κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται για μια περιοχή λοιπόν πολύ επικίνδυνη και δύσκολη για τις δράσεις της UTM. Δύσκολη από το 2014 είναι πλήρως λειτουργική στο Μογκαντήσου η UTM. Αρχικά δραστηριοποιούταν στην Ουγκάντα. Και χάρη στις προσπάθειες των ε, μελών των ε, αντιπροσωπιών μας είχαμε μπορέσει να αποτρέψουμε γεγονότα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο της Γκάρης ε, με πάνω από 100 παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλο κομμάτι δηλαδή της ελίτ της χώρας με ένα τα επίπεδα εκπαίδευσης στην Κένια χάθηκε μια κατάσταση φρικτή και βέβαια περιμένουμε να μας δώσει ο ταξιέρχος την ενημέρωση για την κατάσταση. Η εντολή της UTM παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2016. Θα έχουμε επίσης τον ε, Διευθυντή της ERP Κλόντι ως δεύτερο μιλητή θα έρθει πολύ σύντομα στην αίθουσα δίνω όμω πρώτα το λόγο Όχι, νομίζω θα δώσω το λόγο πρώτα στον ε, ταξιέρχο. Αντώνιο Μάτσι. και όταν έρθει και ο κύριος Σικλόντε θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί και εκείνος και θα επανέλθουμε πάλι στη δική σας παρουσίαση. Εάν συμφωνείτε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Για μένα είναι τιμή η παρουσία μου εδώ για να σας πω δύο λόγια για την αποστολή μας στη Σομαλία. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Η αποστολή μας στη Σομαλία συμπληρώνει πέντε χρόνια φέτος. Καθορίστηκε το 10 σε ανταπόκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να χορηγηθεί βοήθεια και εκπαίδευση στις σομαλικές δυνάμεις. Άρχισε στην Ουγκάντα. Για να δούμε, αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις που άρχισαν στο Μογκαντήσιο και μετά η, Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφαλείας ζήτησε την μεταφορά από το μογκαντίσιο για να οικοδομηθούν δομές άμυνας και να βελτιωθούν οι δυνατότητες των δυνάμεων εκεί. Έχουμε 155 πρόσωπα από 11 χώρες συν τη Σερβία, χώρες μέλη συν τη Σερβία. Η νέα μας εντολή τώρα άρχισε την, πρωταπριλιά του 2015 με σαφή εντολή να βελτιώσουμε τον τομέα της άμυνας με συμβουλές αλλά και να στηρίξουμε και να εκπαιδεύσουμε τον Σομαλικό στρατό. Γι' αυτό οι δραστηριότητες μας είναι τριών ειδών. Εκπαίδευση, όπου στοχεύουμε κατά την 20 αποστολή μας μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 να κάνουμε 20 μαθήματα για 1.200 μαθητάς σε θέματα όπως διοίκηση, στρατιωτική αστυνομία, στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών κλπ. Και χορηγούμε και καθηγητάς για να γίνει μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Επίσης, συμβουλεύουμε τον στρατό της Σομαλίας για να μπορεί να στηρίξει και να βελτιώσει τις υποδομές για την ασφάλεια και την περαιτέρω εκπαίδευση. Οι σύμβουλοι προέρχονται κυρίως από το Υπουργείο Αμήνης με επικεφαλής τον αρχηγό του. Επίσης χορηγούμε τεχνικές συμβουλές σε τομείς όπως διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση υλικών πόρων, σχεδιασμό και πολιτική. Αυτό είναι ουσιώδες για να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες του Σομαλικού στρατού και να αυξηθεί έτσι και η πολιτική εποπιτεία. Μέχρι τώρα έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 μέλη του Σομαλικού στρατού αλλά έχουμε χορηγήσει και υπουργικές συμβουλές και στρατηγικά σχέδια. Όπως είπε πρόσφατα το Υπουργείο Αμήνης της Σομαλίας, η αποστολή μας έπαιξε ουσιαστικό ρόλο για την διασφάλιση του Μογκαντήσιου. Επίσης εξετάζουμε τη δυνατότητα αύξησης της στήριξής μας προς το SNA που λέμε με κεντρική ιδέα να μπορέσουμε να κάνουμε τα προγράμματά μας πιο βιώσιμα. Τώρα μπορεί να ακούγονται αυτά θεωρητικά ακόμα, αλλά ελπίζουμε να καταλήξουν σε κάτι ρεαλιστικό και υλικό με βάση αυτά που ζήτησε το ψήφισμα 1872 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο τον Σομαλικό στρατό, ας πούμε, το στρατιωτικό νοσοκομείο είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες μας. Εκεί θεραπεύονται οι στρατιώτες που έχουν πληγωθεί στα μέτωπα και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν περισσότεροι πόροι για τη στήριξή του. Um, Τώρα για τη σφαιρική προσέγγιση μας. Η αποστολή μας είναι η πρώτη μόνιμη αποστολή στη Σομαλία. Υπάρχει και σαφής δομή διοίκησης. με τη γενική ευθύνη του υπευθύνου της αποστολής. Έχουμε βοηθηθεί και από τις υπηρεσίες του μας στις Βρυξέλλες. Συνεργαζόμαστε με το UMS, EPD, UMC, όλα αυτά. Στη Σομαλία έχουμε επαφές με και με τους πρεσβευτές μας. Το προσωπικό μου δύο φορές το μήνα συνεδριάζει για να συντονίσει και τα τρία τμήματα της αποστολής. Και έχουμε συνδέσεις και με τις υπόλοιπες αποστολές ESDP για να υπάρξουν συνέργειες και συνεργασίες. UTM Somalia is well Εκτός αυτού υπάρχει και συντονισμός γενικά των Ηνωμένων Εθνών παίζουμε σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση του συντονισμού και την συμπροεδρία με τον ΟΗΕ, τα κράτη-μέλη και άλλους προμηθευτάς εκπαίδευσης. Τέλος, νομίζω ότι η αποστολή μας ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στη Σομαλία. Αυτή η τριμερής προσέγγισή μας μας επιτρέπει να λύσουμε τα προβλήματα της Σομαλίας με σωστή διαχείριση σε θεσμικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά η Σομαλία παραμένει σε λεπτή κατάσταση και χρειάζεται ακόμη βοήθεια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες για τη στήριξη των Σομαλικών ενόπλων δυνάμεων. Σας κατευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε ταξίαρχε. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω επισήμως ε, τον ε, κύριο Γκάμπορ Ίκλοντι, τον πρέσβη Γκάμπορ Ίκλοντι, ο οποίος είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού CMPD. Ο κύριος Ίκλοντι συμφώνησε να συζητήσουμε δύο σημεία από κοινού το πρώτο από με τον ταξιάρχο Μάτζη, η κατάσταση Σομαλία. Και το δεύτερο είναι η, γενική ανταλλαγή απόψεων και επισκόπηση των ευρωπαϊκών αποστολών όλες τις πτυχές της και όπου και αν αυτές αναπτύσσονται. Κύριε Κλίντ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι βεβαίως είχα την δυνατότητα να ακούσω τι είπε και ο ταξίαρχος, αλλά ε, θα προσπαθήσω να συμπληρώσω πολύ σύντομα και να εστιάσω στα ερωτήματα που ενδεχομένω να έχετε σε σχέση με την εκπαιδευτική αποστολή και την κατάσταση στη Σομαλία. Γνωρίζετε ίσως ότι η στήριξη για τη σταθεροποίηση Σομαλίας ε, που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και να αναφέρω ότι καταρχάς ε, παρέχουμε τη περισσότερη, το μεγαλύτερο μέρος αναπτυξικής βοήθειας στη Σομαλία, και το ΕΝΙΣΟΜ, αυτή τη μονάδα δηλαδή που ουσιαστικά αναλαμβάνει το κομμάτι το στρατιωτικό, την υποστηρίζουμε. Και έχουμε και τις τρεις αποστολές, Ομαλία, δύο στρατιωτικές, την Αταλάντη, που είναι η μόνη ναυτική επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε, μάλλον αμυγός Ευρωπαϊκή, και έχουμε και την EUTM, την εκπαιδευτική αποστολή. Και την νεότερη, την τρίτη, έχουμε τον Νέστορ για τη δημιουργία μη στρατιωτικών υποδομών. Ποια είναι η ομορφιά αυτής της προσέγγισης. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την επιχείρηση Αταλάντη και τις προσπάθειες καταπολέμησης της πειρατείας. Το ωραίο λοιπόν είναι ότι με τις τρεις αυτές αποστόλες αλλά και με άλλες ε, δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστιάζει μόνο στα συμπτώματα της πειρατείας στη θάλασσα αλλά προσπαθεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει ε, τις βαθιές αιτίες της πειρατείας εξού και οι αποστολές, οι εκπαιδευτικές που συνδυάζουν το στρατιωτικό και το μη στρατιωτικό σκέλος. Συνεργάζονται τα μέλη των δύο αποστολών στη Σομαλία και αυτό συνιστά μείζωνα διαφορά αν συγκρίνει κανείς ε, την ε, επιχείρηση Ocean Shield για παράδειγμα του ΝΑΤΟ ή την Αταλάντη και τις άλλες αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πολιτικής πλευράς, παρά τις ελλείψεις που είναι και προφανείς στη Σομαλία, η χώρα πλέον βρίσκεται σε θετική τροχιά. Βέβαια όλα αυτά είναι και, έχουν και να, να κάνουμε το με ποια χώρα συγκρίνει κανείς τη Σομαλία. Πάντως φαίνεται ότι βγαίνει από την Άβυσσο σιγά σιγά η, η χώρα αυτή, η Σομαλία. Παρά όμως τη σχετική αυτή επιτυχία της Σομαλίας, η κατάσταση της ασφάλειας παραμένει σαφώς ε, ρευστή. Είναι σαφές ότι είναι πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος της ε, προσπάθειας οικοδόμησης κράτους. Αρνητικός αντίκτυπος. Άρα, συνάγω από όλα αυτά ότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής στην Σομαλία είναι πάρα πολύ απαραίτητη. για την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που έχουμε δώσει στη Σομαλία και για να υπάρξει πρόοδος. Υπάρχει πληθώρα ανακών στη Σομαλία. Δεν έχει καν νόημα να κάτσουμε να τις απαριθμίσουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε κυρίως στους τομείς εκείνους όπου μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τις φιλοδοξίες μας, τους πόρους μας θα πρέπει να τους ε, συγχρονίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Για να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια, ορμολογούμε μια νέα διαδικασία. Το PFCA, Political Framework for a Crisis Approach, πολιτικό ναι. πλαίσιο για μια προσέγγιση στην κρίση. Είναι μια συνοπτική αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Πώς ε, έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες όταν θα έχουμε όλο το πλαίσιο που περιλαμβάνει βέβαια και τη δράση άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όχι μόνο στη Σομαλία, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, δεν μιλώ μόνο για την οργανισμούς. Γνωρίζουμε ότι στη Σομαλία γιδίνονται πόλεμοι δια προσώπου. Υπάρχουν ξεκάθαρα συμφέροντα και θα πρέπει να δούμε πού εστιάζουμε με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις μας ε, στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Είναι επιτυχημένες αυτές οι αποστολές. Έχουν οι επενδύσεις απόδοση, οι επενδύσεις των κρατών μελών. Αυτό είναι η δυνατότητά μας λοιπόν και η ευκαιρία που έχουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και εξελίσσεται η κατάσταση όχι μόνο στη χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία που έχουμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και όχι να βλέπουμε ε, μέσα από τη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση και πώς θα είναι στο μέλλον τα πράγματα γύρω στα τέλη του 2016. Οπότε και λίγη η εντολή και η θητή και των τριών αυτών αποστολών. Που λαμβάνουν χώρα εκ Και που όπως σας είπα συγχρονίστηκαν πριν από λίγο καιρό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαγράφεται στο μέλλον η κατάσταση. Να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Και μετά σε αυτό το πλαίσιο θα αξιολογήσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε ήδη αναπτύξει. Για να δούμε αν δίνουν καλά αποτελέσματα, αν δίνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν χρειάζονται βελτιώσεις. Για πρώτη φορά θα γίνει κάτι τέτοιο. Βάσει λοιπόν αυτό το PFCA, αυτό του πολιτικού πλαισίου κτλ. θα ξεκινήσει μια κοινή αξιολόγηση των τριών αποστολών το καλοκαίρι συγκεκριμένα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Οπότε μετά μπορούμε να κάνουμε τι απαραίτητε προσαρμογές. Την προηγούμενη εβδομάδα γυρίσαμε το Ναϊρόμπι, ήμασταν με τον α, ταξίαρχο. USR, ε, αντιπροσωπεία, το γεωγραφικό γραφείο και κάποιοι άλλοι διεθνείς παράγοντες, Ηνωμένα Έθνη, Ένισον, Ευρωπαϊκή Ένωση, mm ΙΠΑ. και συνεδριάσαμε όπως επίσης και με τις τοπικές πρεσβείες Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητήσαμε το πώς βλέπουμε την κατάσταση να εξελίσσεται. Αυτό ήταν ένα είδος ε, έναρξης της όλης διαδικασίας. Το θέμα είναι αν κάνουμε τα σωστά πράγματα και με το σωστό τρόπο. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ως αφετηρία όχι μόνο την κατάσταση στη Σομαλία, αλλά και τα συμφέροντα της Ένωσης. Δηλαδή, σε ό,τι κάνουμε είναι σημαντικό να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και να δίνουμε αποτελέσματα. Ένα από τα συμφέροντά μας βέβαια είναι η περιφερειακή σταθερότητα ή η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οργάνωση Al-Shabaab και η περαιτέρω διάδοση αυτής της υπηρεσίας ε, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να κερδίσει αυτό τον πόλεμο η Ελσαμπάμπ και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να χάσει. Την Έμισομ λοιπόν προσπαθούμε να την ενθαρρύνουμε, είναι αυτοί που πολεμούν επί τόπου και το ίδιο σκοπό έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή άλλα τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες και σε αυτή την ανάγκη την συγκεκριμένη της περιφερικής ασφάλειας, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει με έναν ολοκληρωμένο, συντονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρόπο. Έχουμε και το ναυτικό εμπόριο. Υπάρχουν εδώ ξεκάθαρα συμφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται καν να σας το πω αυτό. Έξω και γίνεται μια συζήτηση για την Αταλάντα, την επιχείρηση Αταλάντη, που ουσιαστικά έπεσε θύμα της επιτυχίας της σε μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως σας γνωρίζετε, δεν υπήρξαν επιτυχημένες ε, απόπειρες πειρατεία στη θάλασσα και εύκολα μπορεί κανείς να καταλήξει το συμπέρασμα ότι ε, ήρθε η ώρα να βγάλει το μηχάνημα από την πρίζα και να σταματήσει στην αποστολή. Μα αν γίνει αυτό όμως θα επανέλθουν πάρα πολύ γρήγορα στην περιοχή οι πειρατές. Θα πρέπει να βρούμε λύση στο πρόβλημα της ε, πειρατείας και στην ξηρά. Αν δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος και από το EUCAP Nestor και από την παιδική αποστολή, και αν δεν έχουμε αποτελέσματα απτά ε, στο πολιτικό επίπεδο, από την εκπαιδευτική αποστολή, θα επανέλθουν οι πειρατές αν αυτά δεν επιτευχθούν στην πτυρά, θα πάνε στη θάλασσα πειρατέ. Ένα από τα συμπεράσματα τη συνάντηση του Ναϊρόμπι ήταν ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την εντολή των αποστολών και να εστιάσουμε σε αυτά που θα μας δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι εκεί, στην περιοχή, η κατάσταση εξελίσσεται, μεταβάλλεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο, ότι είναι η εμένη. Και σε εσωτερικό επίπεδο το συστησαμε πέρυσι, αν δει στο το χάρτη, θα πει, μα ήδη έχουμε κάποιους, ε, κάποια μέσα, κάποιους πόρους και πάει εκεί. Μήπως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα και έκτατες καταστάσεις εκεί. Αντί να είναι πάρα πολύ περιοριστικά, πολύ περιοριστικές οι αποστολές, που δεν δίνουν κανένα περιθώριο, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και να βλέπουμε τι απαιτούν οι καιροί κάθε φορά. Βέβαια πιο εύκολο το λέει κανείς παρά το κάνει. Θα πρέπει να δούμε και τις διαφορές μεταξύ των προσώπων ε, των κρατών μελών. Αλλιώς σκέφτονται τα πράγματα αυτοί που είναι εδώ και αλλιώς αυτοί που είναι στο Ναϊρόμπι. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το δέντρο αλλά και το δάσος λένε εδώ. Υπάρχουν ε, ανταγωνιστικές μεταξύ τους προτεραιότητες. Πολλοί επίσης βλέπουμε εδώ, όταν πάντα ε, κοιτούμε προς την περιοχή, ε, και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους σπόρους, κάτι που μπορεί να μην το βλέπουν εκεί απαραίτητα. Πρέπει όμως να σχεδιάσουμε την εντολή κατά τρόπο τέτοιο ώστε η συμβολή μας στην ασφάλεια της Ομαλίας να είναι πιο σημαντική. Τώρα, σε ό,τι την ίδια την αποστολή, την εκπαιδευτική αποστολή, ο ταξιάρχος ε, Μάτζη ήδη σκιαγράψει τις βασικές δραστηριότητες αυτής της αποστολής που είναι σίγουρα κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης και εγώ θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω μια αλλαγή, μείζον αλλαγή όταν η αποστολή από πολύ, την πολύ ειρηνική Ουγγάντα πέρασε στο Μογκαντίσου, που έχει την έδρα της σήμερα και από όπου ασκεί το συμβουλευτικό ρόλο, παρέχει καθοδήγηση, εκπαίδευση. Και πρόκειται για πραγματική αλλαγή παραδείγματος. Η εντολή της αποστολής εκπνέει στα τέλη του έτους και ήδη είχε ζητηθεί και προηγουμένως ε, να υπάρξει κάποια επεξεργασία αυτής της εντολής και να εστιάσει περισσότερο αποστολή στην παροχή στρατηγικών συμβουλών. Οι αρχές της Σομαλίας επίσης δεν φαίνεται να έχουν ξεκάθαρη αντίληψη για το είδος των ενόπλων δυνάμεων που θα ήθελαν και που θα χρειάζονταν. Δεν έχουν δόγμα. Και είναι πολύ δύσκολο να παρέχει κανείς βοήθεια και εκπαίδευση αν δεν γνωρίζει για ποιο λόγο εκπαιδεύει Γι' αυτό και η εν λόγω δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο της αποστολής. Κατακλείδη. Κάποιες ε, πρόσθετες παρατηρήσεις. Πανακύπτουν και πολύ σχεδόν στις συζητήσεις που έχουμε. Η εκπαίδευσή μας γίνεται για τους σωστούς στόχους. Είναι ένα ερώτημα. όπως οι πρεσβείες τα έλεγαν στη Σομαλία. Βασική ανησυχία και μέλημα είναι να αγωνιστούμε κατά της Al Σαμπάπ. Αυτός είναι ένας στόχος και είναι σημαντικός στόχος, ε, γίνεται, αυτός είναι ο στόχος της αποστολής, αυτό κάνει και ο διοικητής, προσπαθεί να εκπαιδεύσει έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσει και λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης και για να ανταποκριθούμε στην όλο και μεταβαλλόμενη κατάσταση επιτόπου. Επίσης και στο μέλλον μεγάλη σημασία... Α, ναι, Μια ακόμη σκέψη πριν περάσω στο επόμενο σημείο. Η αποστολή έχει την έδρα στο Μογκαντήσου. Σήμερα. Είναι όλο και πιο σημαντικό να μεταφερθεί προς τα έξω εκτός Μογκαντήσου δηλαδή, να κάνει και εκεί, να παρέχει και εκτός Μογκαντήσου εκπαίδευση. Στον Αϊρόπη είπαν, είπαν στρατηγός ότι πρέπει κανείς ε, να παρέχει την εκπαίδευση εκεί που γίνονται και, που και, που γίνονται και εχθροπραξίες. Να περάσεις δηλαδή στην Ήπεθρο, εκεί που είναι το θέατρο των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα προστασία των ε, ε, δυνάμεων, των στρατευμάτων, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα. Με τη βοήθεια βέβαια και της Εμισών και βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει τη χρηματοδότηση. Η στενή αλληλεπίδραση με την Έμισον και στο μέλλον αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τώρα, στον τομέα της εκπαίδευσης, αναρμονισμένες εκπαιδευτικές ε, δράσεις για καλύτερα αποτελέσματα, προστασία δυνάμεων, δηλαδή η έμισο να παρέχει τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες προσανατολισμένες περισσότερο στην καταπολέμηση της al να έχει μια πιο επιθετική ε, στάση, αλλά και να ε, παρέχει προστασία στους εκπαιδευτές εάν ε, μετακινηθούν εκτός Μογκαντήσου, ώστε η χρηματοδότηση μας να πηγαίνει σωστή, σωστή κατεύθυνση. Και επίσης ο εντοπισμός προσωπικού, μάλλον όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού, τι γίνεται, πώς εξασφαλίζεις ότι δεν θα αλλάξουν ε, πλευρά και δεν θα ενταχθούν στην να σε κάποια άλλη ομάδα. Σήμερα που εντοπίστε αποκλειστικά και μόνο στο Μογκαντήσου αυτή η αποστολή, η, τα ενδεχόμενο ελέγχου αυτής της κατάστασης είναι περιορισμένο. Κυρίως πρέπει να βασιστούμε στις τοπικές αρχές αλλά και στην Έμισο, που είναι παρούσα σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Υπάρχουν μέθοδοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Παραδείγματο χάρη. Εισαγωγή ενό βιομετρικού συστήματο για να εντοπίσετε το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί. Εκπαίδευση και εξοπλισμό. Το είπε και ο ταξίαρχο. Δεν θέλω να επισέλθω σε άχρηστες ίσως λεπτομέρειες. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, Train and Equip, εκπαίδευση και εξοπλισμός, γιατί είναι ο κρίκος που συνδέει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη. Γιατί χρησιμοποιεί τις, ε, τα, τα ισχυρά σημεία στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Είναι η λεγόμενη γενική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση. Μαζί με το Μαλί, η Σομαλία ήταν ένα από τα θέατρα όπου γίνονταν κάποια πιλωτικά προγράμματα τους τελευταίους μήνες με στόχο και η εκπαιδευτική αποστολή της Ένωσης αλλά και άλλες επιχειρήσεις και αποστολές ε, γι' αυτό δραστηριοποιούνται εκεί να αξιολογηθούν οι ανάγκες, τι εξοπλισμό χρειάζονται δηλαδή ένας άλλος στόχος η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων των χορηγών, των χρηματοδοτών, όχι μόνο τα κρατημέλη της Ένωσης και άλλοι, η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Τι δραστηριότητες ε, βλέπουμε από πλευράς χορηγών, χρηματοδοτών. Και τρίτον, εκτίμηση, αξιολόγηση κινδύνων με την παροχή του εξοπλισμού. Τι εγγύησεις έχουμε ότι ο εξοπλισμός ο παρεχόμενος δεν θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για σκοπούς ασύμβατους με τους στόχους της Ένωσης. Για να είμαι σαφής, δεν μιλάμε για φωνικά ε, όπλα, για φωνικό εξοπλισμό. Αυτό είναι εθνικό, εθνική απόφαση. Αν ένα κράτος μέλος ή ένα μη κράτος μέλος αποφασίσει να παράσχει πυρομαχικά εξοπλισμό στη Σομαλία, μπορεί να το κάνει δεν είναι ευθύνη της Ένωσης, δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης και δεν χρηματοδοτείται από τον ενωσιακό προεπλογισμό για να είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα εδώ είναι, και ανήκω παρέθεση εδώ, ότι το Training Equip, εκπαίδευση και εξοπλισμός, έχει ως στόχο να εντοπίσει τα βασικά κενά στις προσπάθειες Ένωση να δημιουργήσει ικανότητες και δυνατότητες στις χώρες εταίρους. Το κενό αυτό είναι συνέπεια του σχεδιασμού των χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων που έχουμε. Η απόφαση επίσης για το πώς θα ερμηνεύσουμε τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει ρόλο. Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε πολύ ξεκάθαρα ότι μια στρατιωτική οργάνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τίποτα ούτε και για μολύβια, αν είναι στρατιωτική οργάνωση. Αν υπάρχουν ερμηνείες που δεν εμπίπτουν ε, σε αυτά τα που μπορεί να χρηματοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία. Η ερμηνεία της Κομισιόν είναι αυτή, έτσι. Και υπάρχει και η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι, λάθος. Ε, είπα, λένε ότι με βάση το άρθρο 41.2 της συνθήκης, ως έχει αυτή τη στιγμή, και με βάση το διατάξει των χρηματοδοτικών μηχανισμών κανονισμών, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την στήριξη αυτών των στόχων δημιουργίας υποδομών και ικανοτήτων. Γίνεται συνεχώς ε, μια συζήτηση για αυτό το πρόγραμμα Train and Equip που θα είναι ίσως και το σημαντικότερο ε, αποτέλεσμα που θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Θα συνεδριάσει σύντομα και ίσως υπάρξει κάποια όθηση για να μπορέσει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα να κλείσει. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση. Ακόμη και αν κάνει η δημιουργία αποδομών η Ένωση παντού, γιατί αυτή είναι η ουσία, η δημιουργία κρατών, οικοδόμηση κρατών που θα μπορούν να λειτουργούν σωστά. Αν αφήσουμε έξω το σκέλος ε, της άμυνας, δεν θα μπορέσει η εκάστοτε χώρα να ε, είναι σταθερή, βιώσιμη, να λειτουργεί. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, η λόγω χώρα μπορεί να καταρρεύσει και αυτό να οδηγήσει σε κίνδυνο για όλες τις άλλες επενδύσεις που θα έχουν γίνει σε άλλους τομείς στη χώρα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαψη κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή δημιουργία υποδομών, capacity building εν γέννη, ε, παντού. Και είναι κάτι που κερδίζει έδαφος και στη, στο στρατιωτικό και στο μη στρατιωτικό σκέλος. Αυτά για την εκπαίδευση εξοπλισμού. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι όταν το Συμβουλίο πάρει τις αποφάσεις του τον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα, και μπορεί κάποιες λύσεις να ξεκινήσουν μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς μας πλαισίου. Είναι σημαντικό σε αυτά τα θέατρα τουλάχιστον όπως είναι το Μαλή Σομαλία να ξεκινήσουν έστω και περιορισμένα προγράμματα εξοπλισμού. Αυτό είναι σημαντικό. Και μια τελευταία λέξη. Λοιπόν, αυτό είπα πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή συνδυασμό εκπαίδευση με εξοπλισμό, γιατί λίγη είναι αξία της εκπαίδευση αν δεν υπάρχει εξοπλισμό για να μπορέσουν να φέρουν πέρα στα καθήκοντά τους οι εκπαιδευόμενοι οι Και επίσης θα πρέπει να είναι σταθερή η προσπάθεια, να διατηρηθεί. Και εδώ παίζουν και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν. Πάντα φέρνω το παράδειγμα του Αφγανιστάν. 250.000 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν, άφησαν εξοπλισμό πίσω. Αν δηλαδή η προσπάθεια δεν διατηρηθεί, δεν είναι σταθερή, ο εξοπλισμός ε, υψηλής τεχνολογίας ή όχι, ε, θα χρησιμοποιείται μέχρι να διαλυθεί ή να χαλάσει. Και όπως είπε και ένας συνάδελφος, βλέπει νεκροταφεία εξοπλισμού εποχής ε, σοβιετικής, σοβιετικού τύπου να σαπίζουν στην περιοχή εκεί. Άρα μόνο αν είναι μια σταθερή προσπάθεια, αν είναι βιώσιμη προσπάθεια, δεν θα έχουμε νέα τέτοια νεκροταφεία. Και δεν θα βρούμε εκεί να σαπίζουν και αμερικανικός και ευρωπαϊκός εξοπλισμός και όπλα. Οι σχέσεις με τις άλλες δύο αποστολές τώρα, ε, όπως το είπε και ο ταξίαρχος, είναι πολύ σημαντικές, θέλουμε να δώσουν αποτελέσματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέτρα ε, της Επιτροπής. θα ε, σταματήσω όμως εδώ γιατί μακρηγόρησα. Όχι, όχι, δεν ήταν ε, μακροσκελής η ομιλία σας, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους και τους συνεργάτες τους ότι έχουμε και ένα κομμάτι συνεδρίασης για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες και τις δυνατότητες τους που προβλέπεται στις 28, δεν απατώμε, Μαΐου. αλλά και σήμερα. Κατά την συζήτηση με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου θα έχουμε την ευκαιρία, έστω και εν μέρη, να το συζητήσουμε. Ας αρχίσει η συζήτηση λοιπόν με τον κύριο Γκάλερ πρώτα. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσαν να είμαι παρόν από την αρχή. Ενημερώθηκα όμως για τα όσα υπόθηκαν. Η κατάσταση της ασφάλειας ορισμένα σημεία της Σομαλίας αναπτύσσεται κατά τρόπο όχι θετικό, όπως βλέπουμε και από επιθέσεις και στην πρωτεύουσα, αλλά και με την επίθεση βάρους ε, του αυτοκινητών εθνών με 7 τουλάχιστον νεκρούς. Υπάρχουν όμως αναφορές ακόμη και για 10 από το BBC. Η Αλσομπάπ φαίνεται ότι έχει την ευθύνη και ότι είχε αποσυρθεί προς τα βόρεια της χώρας. Δεν έχει σταθεροποιηθεί λοιπόν η χώρα όπως περιμέναμε. για τον ε, ταξίαρχο Μάτζη αλλά και για τον κύριο Ικλόντε λέτε ότι πρέπει να υπάρχει το δυναμικό ως διάθεση. Βεβαίως, το στρατιωτικός εξοπλισμός ήταν ούτως ή άλλως ε, απειρχαιωμένος εξοπλισμός που είχαν διαθέσει τα κρατημέλη. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι. Και αν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης νέου εξοπλισμού κατά τρόπο συντονισμένο μεταξύ των κρατών μελών. κατά τρόπο αλλά και να είναι κατάλληλος ο εξοπλισμός. Επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε το τι είναι δυνατόν, δυνάμει του άρθρου 41 δεύτερη παράγραφος συνθήκης, με την πιο ευέλικτη, εναλλακτική, δηλαδή να κοιτάξουμε τι γίνεται πριν από τη στρατιωτική επέμβαση, αλλά και μετά από μια στρατιωτική επέμβαση, κατάρτιση, εκπαίδευση, προετοιμασία, και βέβαια σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαμε εδώ έχουμε να κάνουμε τα βασικά στοιχεία οικοδόμησης κράτους σε αυτήν την κατάσταση. Με αντίπαλο την Ανσαμπάπ. Άρα θα χρειαστεί οπωσδήποτε αυτή η διάσταση, αυτό το μέσο του εξοπλισμού του Ρωτικού. Μια άλλη ερώτηση για τον κύριο Ικλόντι. Ε, ενημερώθηκα ότι κάνατε ερωτήσεις αν κάνουμε το σωστό και αν κάνουμε το σωστό με το σωστό τρόπο. Περιμένω να μας δώσετε εσείς τις απαντήσεις σε αυτές τα ερωτήματα. Θα πρέπει και η Επιτροπή να έχει τις απαντήσεις, διάθεση τις σωστές απαντήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε με την περίπτωση της ε, Σομαλίας και την καλύτερη ε, συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, παραδείγματι για την αμισόν και χρηματοδότηση από το Αφρικανικό Κονδύλιο Αφρικανικών Μέσων. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να μας πείτε περισσότερο για τις ανάγκες της ε, χρηματοδότησης αμισόν. Ευχαριστώ, Ζιλ Παρνιού, σοσιαλιστές. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν πληρέστατες. Ταυτόχρονα γερνούν πολλά ερωτηματικά. Έχουμε να κάνουμε μια χώρα που βρίσκεται από το 1991, από τις 26 Ιανουαρίου του 1991 σε εμφύλιο. Κοινή επέμβαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένωσης μαζί με την ε, UTM και η παρέμβαση της Amazon με το Ηνωμένα Έθνη που προηγείται γράφονται μέσα σε μια κατάσταση παράδοξη καθώς από το 2011 τουλάχιστον το σύνολο των στρατιωτικών δράσεων κατά των στασιαστών, των Ισλαμιστών στασιαστών της Al-Shabaab βασικά οδηγούν σε οπισθοδρόμηση αυτές τις Ισλαμιστικές ομάδες. Έφνης όμως βλέπουμε τον Απρίλιο την επανεμφάνιση μιας σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων, όχι μόνο στη Σομαλία, αλλά και στις γύρω περιοχές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. η αποτελεσματικότητα στρατιωτική με την επιτόπου δράση το τελευταίο διάστημα θεωρείται ότι δεν έφερε τους αναμενόμενους καρπούς. Μια και έχουμε αντιμετωπίσει την al που βρίσκεται εκτός Σομαλίας ή, και, ή στα βόρεια όπως έλεγε ο συνάδελφος ή και αλλού και εν πάση περιπτώσει μήπως τελικά δεν κάνουμε αυτό που χρειαζόταν σε σχέση με τις επιλεγήσεις από αυτούς ε, δραστηριότητες και τις τοποθεσίες για τις δραστηριότητες. Και επίσης, ε, όπως και, ε, όπως και η πρόεδρος και άλλοι συνάδελφοι της Επιτροπής, ήμασταν σε μια αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου διαπιστώσαμε πόσο ακαθόδης είναι η σχέση μεταξύ των δυνάμεων του ΟΗΕ και του τοπικού πληθυσμού της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Στη Σομαλία τι γίνεται. Εκεί έχουμε παρουσία της Αμισόμ. Υπάρχει λοιπόν αντίστοιχα ακανθώδης κατάσταση, δύσκολη κατάσταση όπως είχαμε διαπιστώσει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η Πρόεδρος, κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που με ανησυχούν σοβαρά βασικά ζητήματα. Είπατε ναι. ότι η Σομαλική κυβέρνηση δεν ξέρει τι στρατό θέλει. Ναι. Άρα ερωτώ. Εμείς τι στρατό εκπαιδεύουμε. Για ποιο λόγο. Γιατί αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει πόλεμος. Και η Αλσαμπάπ το έχει καταλάβει πολύ καλά αυτό. Άρα όταν ένας εχθρός ε, έχει καταλάβει πολύ καλά μια κατάσταση, εμείς ε, παραμένουμε άναυδοι ακούγοντας ε, ότι οι παράγοντες, τέλο πάντων ε, η ε, σομαλική κυβέρνηση που είναι κάτι πιο φιλοσοφικό παρά πραγματικό δεν ξέρει τι θέλει. Άρα η εκπαιδευτική αποστολή αυτά που κάνει και ξοδεύει είναι τα αντίστοιχα με αυτό που κάνει στο Μαλί. Εγώ πηγαίνοντας ε, με μια αποστολή που όλοι λένε ότι ήταν πολύ επιτυχημένη στο Μαλί, όταν γύρισα έμεινα άναυδος. Πρώτη ερώτηση. Γίνεται παθητική εκπαίδευση που είναι ε, τελείως γελίο. Ε, μιλάω για το στρατό το σομαλικό, κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στο Μαλί. Κάποιος στρατιωτικός πρέπει να μου εξηγήσει τι θα πει αμυντική ε, εκπαίδευση στην έρημο. Μπορεί κάποιο να μου το εξηγήσει. Επίση, ε, παρέχεται ο κατάλληλο εξοπλισμό ή αυτό εξαρτάται από τη σομαλική κυβέρνηση όπω και από την κυβέρνηση του Μαλή. Άρα δεν υπάρχει εξοπλισμό. Άρα πώς υπάρχει εκπαίδευση χωρίς ε, εξοπλισμό. Τρίτη ερώτηση που μπαίνει έτσι και λίγο ε, στη σφαίρα του αστείου, χιουμοριστική πλέον αν εκπαιδεύουμε το στρατό της Σομαλίας όπως το Μαλί ε, στον ποταμό, ενώ δεν υπάρχει στη Σαχάρα ποταμός, ε, τι κάνουμε ακριβώς, ε, είναι αστείο. Και τέταρτον, τι στρατολόγηση γίνεται στη Σομαλία που είναι το μόνο ομοιογενές εθνικός κράτος που όμως έχει, χωρίζεται σε φρατρίες οι οποίες μισιούνται. αυτοί που στέλνουν οι λεγόμενες πολιτικές ομάδες ουσιαστικά είναι ομάδες που έχουν ε, τη δύναμη επιτόπου αυτοί στέλνουν, ε, αυτοί στρατολογούν ή γίνεται μια ολοκληρωμένη ομογενής ε, στρατολόγηση και είναι αυτό βιώσιμο. Έχουμε τους Νταρότ, τους Χίτε, τους Μουσαχεντίνου και άλλες φρατρίες που υπάρχουν στη Σομαλία. Και Τέταρτο. Όταν τελειώνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ε, θέλουμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Εδώ ας πούμε ότι έχουμε 11 παίκτες, χωρίς να ξέρει κανείς την τακτική που ακολουθούν και δεν ξέρουμε και τι κάνουν στο γήπεδο των εισαγωγικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Ε, δεν μπορεί να βασίζονται στα ξένα στρατεύματα τα αφρικανικά και ευρωπαϊκά στρατεύματα, εντάξει δεν κάνουν πόλεμο τα ευρωπαϊκά και όταν ε, γίνεται αυτό από τα αφρικανικά δημιουργούνται εσωτερικά μίση πολύ βαθιά. Έχουμε τους σύφτας, ε, τους, ε, αυτές τις συμμορίες στη, στην Κένια αυτά τα αφρικανικά στρατεύματα πώς γίνονται αποδεκτά σε ομαλή από ένα πληθυσμό που ιστορικά έχει αντιπαραθέσεις με τη γειτονική χώρα Κένια. Πέρα λοιπόν ε, της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, ε, πραγματικά και σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό πώς μπορούν να είναι αποτελεσματικοί αυτοί που εκπαιδεύουμε και έπειτα. Τι γίνεται με αυτούς που εκπαιδεύουμε, αυτές τις δυνάμεις. Ε, πληρώνονται από Λιποτακτούν, τι κάνουν ακριβώς. Γιατί αλλιώς ε, θα τρέχουν να φύγουν μόνο στο άκουσμα ότι πλησιάζει ο εχθρός, όχι να τον βλέπουν. Και έπεται για την πειρατεία και την καταπολέμηση της πειρατείας που είναι σίγουρα πολύ ε, σημαντικό να καταπολεμηθεί. Οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, καμία δυνατότητα επιβίωσης για τους αλείς, όσο η διεθνής κοινότητα επέτρεπε το σφετερισμό των ελευτικών πόρων ή να πέφτουν, να διατίθενται στις ακτές της Σομαλίας, ε, να απορρίπτονται χημικά προϊόντα, κάτι αποτρόπαιο. Ωραία, να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, αλλά επιτρέπουμε και μια αναλλακτική οικονομική δραστηριότητα. Και για να τελειώσει ένας πόλεμος γίνεται ένας πόλεμος άλλος. Εμείς τι πόλεμο κάνουμε πέραν του διοικητικού. Αυτή είναι η ερώτηση τελευταία. Thank you. Mrs. please. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ για τις αναλύσεις και τις ερωτήσεις. Μακάρι να, μπορούσαμε να κοιτάξουμε στην κρυστάλλινη σφαίρα για να δούμε τι θα μας φέρει το μέλλον. για τον ε, στρατηγό Μάτζη. Πώς αξιολογείται τη στρατηγική, τις στρατιωτικές εξελίξεις, στρατιωτική κατάσταση στο μέλλον. Γιατί υπάρχουν ε, εκτιμήσεις ότι από το International Crisis Group ιδιαίτερως ότι μπορεί αυτές οι αντιπαραθέσεις με τα al να χρονίσουν. Έχετε κάποια εκτίμηση εσείς? Και επίσης, στην προηγούμενη θητεία είχαμε συστήσει αρκετές φορές τον εξή τομέα για την ε, επιστράτευση παιδιών ο στρατιωτών. Είχαμε δει και από τις εφημερίδες και από, τις, ε, από τα τηλεοπτικά κανάλια σαφείς αναφορές και είχε ενημερώσει ο Οργανισμός Εθνών ότι στρατιολογούνται παιδιά Και αυτό μπορεί να ήταν κάτι που αφορούσε τη μεταβατική κυβέρνηση της Σομαλίας, αλλά θα πρέπει να δούμε εμείς αν εκπαιδεύουμε στρατιωτικές δυνάμεις Σομαλίας, ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει εγερθεί ήδη σε σχέση με τη Σομαλία. Και τότε η απάντηση που είχαμε λάβει ήταν ότι την κατάσταση την παρακολουθούν. Ερωτώ λοιπόν, γίνεται τίποτε, έχει γίνει τίποτε, υπάρχει κάποια αποτελεσματική και αξιόπιστη δράση για την αντιμετώπιση της στρατολόγησης παιδιών στρατιωτών. Και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Ικλόντι που την έφυξε πρώτος. Οι λιποτάκτες. Το έχουμε ξαναδεί σε, στρα... σε περιπτώσεις στρατιωτικών εκπαιδεύσεων σε διάφορες περιοχές να εκπαιδεύονται στρατιώτες οι οποίοι μετά παίρνουν στο αντίπαλο στρατόπεδο και αξιοποιούν τις δυνατότητες ε, και το δυναμικό που έχουν λάβει. Υπάρχει λοιπόν κάποια αξιολόγηση του πόσοι από αυτούς ε, τους λιποτάκτες έχουν περάσει στην Αλσαβάπ ή έστω εκτίμηση δική σας. Και για τον κύριο Ικλόντι που λέει ότι οι εξελίξεις είναι θετικές, βλέπετε κάποια πιθανότητα να προχωρήσουν σε μια συνθήκη ειρήνης ή έστω σε ανακοχή στη Σομαλία. Και δεν θα ε, ε, δεν θα διστάσω να διατυπώσω και την άλλη την ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό. Ξέρετε ότι η ομάδα μου ε, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να διτηθέται στρατιωτικό εξοπλισμός. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πιο ανοιχτά. Δεν είναι δυνατόν η παράδοση όπλων να εξαρτάται από κάποια ερμηνεία. Πρέπει να υπάρχει κάποια νομικά δεσμευτική διάταξη, έστω και αν δεν μου αρέσει όποια είναι αυτή, αλλά μια διάταξη η οποία θα επιτρέπει και στον πολίτη να ξέρει τι συμβαίνει και βέβαια τι ε, χρήση ε, έχει ο φόρος τον οποίο καταβάλει. αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με άλλα πιο γενικά ζητήματα όπως τη γενική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχέση με τις παραδόσεις οπλισμών. Λέτε ναι, τα θέματα αυτά των εξοπλισμών είναι ζητήματα των κρατών μελών, όχι της Ένωσης, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι κάτι το οποίο ζητούν οι πλευρές. Και εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο αυτή την κοινή θέση. Άρα η κατάσταση παρουσιάζει αντιφάσεις και θα ήθελα να μου δώσετε εσείς τη δική σας ε, εντύπωση. Ευχαριστώ, Στέτινα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, ταξιάρχο και τον διευθυντή. Να κάνω μια ερώτηση. Το 1993 ναι. Εγώ πέρασα αρκετές εβδομάδες στη Σομαλία, όταν υπήρχε λοιμός με γιώτα. Και εκεί είχαμε ε, ταυτόχρονα εμφύλιο πόλεμο. Δεν βλέπω συσχετισμό των δύο. Αν ε, δεν υπήρχε εμφύλιος πόλεμος δεν θα υπήρχε πείνα και αν δεν υπήρχε πείνα δεν θα υπήρχε εμφύλιος. Και αυτά τα βλέπουμε τα συμπτώματα και σε άλλες ε, περιοχές. Στο Σουδάν για παράδειγμα, στο Νότιο Σουδάν. Και αυτό που λέει σχέση με την ερώτηση που θέλω να σας κάνω, να σας υπενθυμίσω. Ε, αυτό που είπατε για τους ε, λιποτάκτες. Ξέρουμε ότι στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, οι λιποτάκτες που έχουν εκπαιδευτεί δημιουργούν πρόβλημα και αυτό μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση της Σομαλίας. Ουσιαστικά ε, μπορεί, μπορούσαν να λικοτακτήσουν γιατί τους δίνανε ένα σακούλι αλεύρι που δεν μπορούσε να τους δώσει μια άλλη ομάδα. Ε, μήπως μπορεί να γίνει το ίδιο και στην περίπτωση αυτή. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο. Ευχαριστούμε κύριε Ταξίαρχε για την προσέλευσή σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε για τις δραστηριότητες σας λόγω τη στρατηγική σημασία που έχει το κέρας της Αφρικής και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία παραδοσιακά ήταν πολύ δύσκολη χώρα, δηλαδή διακυβερνούνταν δύσκολα Νομίζω ότι κάνετε κάτι πολύ σημαντικό και το εκτιμούμε όλος ιδιαιτέρως όλος. Ο κ. Κλόντης είπε στην εισαγωγή του η Σομαλία βρίσκεται σε θετική τροχιά. Πόσο βιώσιμη είναι όμως αυτή η τροχιά. Γιατί για μένα αυτό που είπατε ήταν τολμηρό. Χαίρομαι ε, αν είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ήσασταν υπεραισιόδοξος. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μήπως μπορούσατε να μας το σχολιάσετε λίγο παραπάνω. Και ένα ερώτημα, σε τέτοιες περιοχές οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής ας πούμε όπως η Κένια Κάποτε το κοινοβούλιο της Ομαλίας έδρευε στο Ναϊρόμπι, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι σχέσεις με την Αιθιοπία, που παίζει και αυτή τελευταία σημαντικό ρόλο. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς είναι, ευχαριστώ. Τώρα οι καλεσμένοι μας να απαντήσουν στα σχόλια που έγιναν. Ο κύριος Ικλάουντι πρώτος και μετά ο ταξίαρχος Μάγη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Μέχρι αύριο θα μπορούσαμε να απαντάμε. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε όλες. Ελπίζω να μπορέσει ο ταξίαρχος να απαντήσει ορισμένες. Θα αρχίσω και θα δω μέχρι πού θα φτάσω. Θα απαιτούνταν για απάντηση πλήρη βέβαια περισσότερες γνώσεις από ό,τι διαθέτω. Ας αρχίσω όμως και βλέπουμε. Πρώτον, η χορήγηση υλικού. Ο ταξιάρχος θα σας τα πει αυτά, αλλά εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι και στη Σομαλία και αλλού, γιατί και στο Μαλί λέγανε τέτοια, είδαμε ότι και το βασικότερο υλικό λείπει. Μιλάμε για στρατιώτες που εκπαιδεύονται με σορτάκια. Δεν έχουν μπότες, δεν έχουν αρβίλες, δεν έχουν αντίσκηνα. Βασικά πράγματα δεν έχουν. Δεν μιλάμε εδώ για υλικό πολύ πλοκό. και, αλλά βασικό υλικό, να μια στολίτσα. Για να έχουν το αίσθημα ότι σε κάτι ανήκουν. Πρόσφατα κάναμε μια συζήτηση με τον Τεύκο και εδώ θα μπορούσαν όχι μόνο τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Κομισιόν αλλά δίνονται και άλλες ευκαιρίες παραδείγματος χάρη λείπουν οι αρβίλες να ζητήσουμε από τοπικούς παπουτσίδες να τις κάνουν. Έτσι θα έχουν και αυτή η δουλειά. Πολλά τα ωφέλη. Φυσικά δεν μιλάμε για όπλα εδώ αλλά για πολύ βασικά υλικά, βασικό υλικό που χρειάζονται. Επαναλαμβάνω ότι ο ταξίαρχος θα τα πει αυτά πληρέστερα. αλλά και το, πρόγραμμα, το πιλωτικό πρόγραμμα είχε κάνει έναν πρώτο κατάλογο των αναγκών. Βασικό κατάλογο, ρε, βασικό. Βασικό, σύντομο. Όχι τι θα χρειαζόμασταν αν είχαμε όσα λεφτά θέλαμε, αλλά τις βασικότερες ανάγκες. Για το άρθρο 41 και την ελαστικότερη ερμηνεία, ναι, και συμφωνώ θα ήταν η πιο καλή λύση. Θα σημαίνει όμως ότι η δαπάνηση ενωσιακών χρημάτων θα ελεγχόταν. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι η χρησιμοποίηση χρημάτων και από άλλα εργαλεία υπόρους θα κατέληγαν σε υπερβολικά ψηλά δαπάνες. Όχι, όχι. Τώρα αν δεν υπάρξει συμφωνία για πιο ελαστική ερμηνεία του 41-2 και τον μηχανισμό που προϋποθέτει, τότε πιθανότατα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό δημοσιονομικό εργαλείο για τη στήριξη της εκπαίδευσης. Το θέμα είναι ότι το μήνυμα προς τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες τότε να το χρηματοδοτήσετε μόνοι σας. Δεν είναι η σωστή απάντηση αυτή. Φυσικά θα υπάρξουν κατηγορίες υλικού που δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν παρά μόνο από τα κράτη-μέλη. Τα όπλα ιδίω. Τα μικρά εννοείται όπλα. Τώρα για το κατά πόσο κάνουμε το σωστό και το κάνουμε και σωστά το σωστό. Αυτό είναι ακριβώς ο στόχος της αναθεώρησης που θέλουμε να κάνουμε. Αυτός είναι. Έχουν γίνει προσαρμογές και στη δική μας αποστολή και μας αποστολή γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα και σας είπα από πριν ότι τώρα επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ειδικευμένη εκπαίδευση όχι μόνο στη βασική, μέρα, από τη βασική και συμβουλεύουμε και τις τοπικές αρχές αλλά πρέπει να το προσέξουμε αυτό όλος ιδιαίτερος, όλος. Πρέπει δηλαδή το όλο πλαίσιο να το εξετάσουμε πολύ συνοπτικά και μετά να δούμε αν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η Σομαλία σε δύο χρόνια ας πούμε και μετά να δούμε με τι προγράμματα θα σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Ποιοι είναι οι τομείς όπου μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να επικεντρωθούμε σε αυτά. Now the, uh, uh, in terms of, uh, of where financing can come from and um, the African peace. Η Αφρικανική ειρηνευτική διευκόλυνση αραφέστηκε. Με αυτό το θέμα το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο περιφερειακά, όχι εθνικά προγράμματα και γι' αυτό προσπαθήσαμε κι εμείς να εκμεταλλευτούμε τέτοιους πόρους, αυτούς τους πόρους. Αλλά ο τρόπος, ο τρόπος με τον οποίο έχουν συλληφθεί αυτά τα εργαλεία δεν επιτρέπει πάντοτε να τα εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε. Τώρα αν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και αυτά θα τα ξαναπεί ο ταξίαρχος καλύτερα γιατί εκείνο ξέρει τι θέλουμε ξέρει. Θα μας πει εκείνος. Εκείνος. Αυτός. Τώρα ο, τα ΟΗΕ και η Ένωση πώς συνδυάζονται επί τόπου εκεί πέρα, πώς συνεργάζονται. Δεν ξέρω ακριβώς Ποιες είναι οι αρνητικές εμπειρίες από την κεντροαφρικανική δημοκρατία που, που, που αναφέρατε ή που ακούσατε ή που είδατε ή που ζήσατε. Για την κεντροαφρικανική δημοκρατία θα πούμε περισσότερα στον επόμενο γύρο ο ΙΕ θεωρεί τη συνεργασία με την ενωσιακή αποστολή ως υποδειγματική, ως πρότυπο για το μέλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Α, ναι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Πώς τα βλέπει ο κόσμος. Εδώ έχω μόνο δύο εμπειρίες που μου φάνηκαν πολύ θετικές, επιτόπου εννοώ. Αλλά τώρα με την άφηξη, την άρχη της νέας αποστολής, της αποστολής Ιουμάμ, νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Ιουμάμ. Πώς, πώς, Δεν είναι ενωσιακή η επιχείρηση το θέμα μου, είναι για τον της ρώτησα. Πώς βλέπει ο κόσμος στην Κεντρική Αφρική τις δυνάμεις του ΙΕ, του ΙΕ, όχι για την ΟΜΑΜ. Α, ναι, καλό ερώτημα, καλό. Αλλά δεν το ξέρω, δεν ξέρω την απάντηση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ικανοποιητικά. Θα το ελέγξω όμως και θα, και θα το ελέγξω. το τι είδου εκπαίδευση, τι είδου δυνάμει, αυτά θα τα πει εκείνο πάλι, αυτός και τι προσλήψεις γίνονται. Α, η Αταλάντη, μάλιστα. Η Αταλάντη δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το WFP καταρχάς κατά την αντιπειρατική δηλαδή δραστηριότητα, αλλά έχει και άλλα καθήκοντα δευτερεύοντα, και άλλα. Έχει και άλλα. Και την περασμένη εβδομάδα στον Αϊρόμπι τα λέγαμε αυτά με την ε, αντιπροσωπεία της Ένωσης και προσπαθούσαν να μας πούν ότι ίσως αυτές οι ε, αυτά τα δευτερεύοντα καθήκοντα να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη και στο μέλλον θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γίνουν κύρια καθήκοντα, να είναι πιο αντιδραστική, διαδραστική η Αταλάντη, ώστε να μπορεί να αντιδράει γρηγορότερα προς τις, να αποκρίνεται καλύτερα προς τις τοπικές ανάγκες. Είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος των ετοιμάτων και από τις τοπικές αρχές. Κυρίως λένε ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα η Αταλάντη. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα ελαστικότητας και απ' την άλλη πρέπει να γίνει μια σαφής ταύτιση των ενωσιακών συμφερόντων του τομείς δηλαδή όπου μπορούμε να στηρίξουμε με νόημα. Και αυτό θα γίνει μέσα στην αναθεώρηση του καλοκαιριού. Πόσο θα κρατήσει η διαμάχη με τους Σεμπάμπ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν έχω μαντικές ικανότητες. Υπάρχουν πολλές απειλές. Θυμάστε ότι και τον Μπόκο Χαράμ είχε υποσχεθεί να βοηθήσει την Άισις. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Μπορεί και οι Σεμπάμπ να κάνουν το ίδιο. Το ίδιο. Ακόμα κι αν εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις διαφορετικές τρομοκρατικές ομάδες και περιφέρειες που καμιά φορά δεν συνεργάζονται ένα οι πραγματικότητες μπορεί να είναι διαφορετικές επί τόπου μπορεί να υπάρξουν περισσότερες διασυνδέσεις μεταξύ τους δεν αποκλείεται αυτό και αυτό θα μας τα δυσκολέψει τα πράγματα πολύ. Επίσης η λιποτάκτε πράγματι όποτε γίνεται εκπαίδευση δυνάμεων τίθεται και το πρόβλημα της λιποταξίας. Στο Αφγανιστάν ας πούμε έτσι έγινε και καμιά φορά σε πολύ ψηλά ποσοστά. Δεν μπορώ ούτε, δεν τολμώ ούτε καν να τα υπολογίσω τα ποσοστά λιποταξίας μεταξύ των εκπαιδευομένων από την αποστολή μας στη Σομαλία. Υπάρχουν τρόποι να έχουμε καλύτερη γνώση και κατανόηση του προβλήματος, αλλά είπαμε και πριν το βιομετρικά συστήματα, περισσότερη στήριξη από την άμυσον, περισσότερη παρατήρηση, όλα ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Ό,τι. Mm-hmm. οι πιθανότητες ανακοχής και κεχηρίας δεν φαίνονται πολύ πιθανό αυτό γιατί οι σεμπάμπ φαίνονται ότι έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα και ανθίστανται και δεν θα υποχωρήσουν σύντομα. Θα συνεχίσει η διαμάχη λοιπόν. I'll pass the <laughs> floor to you in the meantime. I'm reviewing the further questions. General, please, floor is yours. Ορίστε κύριε Ταξιάρχα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς η ΕΤΕΜ δεν είναι στρατιωτική <laughs> αποστολή. Στόχος μας δεν είναι στρατιωτικός, αλλά να καταρτήσουμε τις στρατικές δυνάμεις να προσφέρουν συμβουλές στους πολιτικούς και στρατηγικούς φορείς του Υπουργείου Αμήνης και τις δυνάμεις του. Αναπτύσσουμε μία μακροπρόθεσμη ε, ικανότητα για το δυναμικό της άμυνας που θα μπορέσει να αποτελέσει τη δυναμή αποτροπή στο μέλλον. καιρό το 2010 κάναμε βασική κατάρτιση, τώρα πάμε σε πιο εξειδικευμένη και κυρίως στριφόμαστε προς την ηγεσία. Επίσης μιλούμε για θέματα θεπών δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων. Συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία υποστήριξης της άμυσων των Εθνών για να καταθέσουμε και μια σειρά εγχειριδίων για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα σε σχέση με τα παιδιά που στρατολογούνται. Πρόσφατα εκδόθηκε διαταγή να απαγορευθεί η στρατολόγηση παιδιών στρατιωτικές ενόπλες δυνάμεις και την αποτροπή της χρήσης παιδιών σε κάθε τομέα δραστηριότητας των στρατιωτικών δυνάμεων σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην οποία έχει προσχωρήσει και η Σωματεία. Αυτό κάνουμε και στο στρατόπεδο Τζαζίρετζο. Είναι κομμάτι δηλαδή του τρόπου με τον οποίο εξηγούμε στου όμορφους την κατάσταση για την κατάρτιση τώρα. Το εξοπλισμό κατάρτισης. Είναι ύψης της σημασίας να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τον εξοπλισμό για την κατάρτιση που χρειάζεται. Ανάλογα με την περίπτωση, Τώρα μιλούμε δηλαδή για θέματα διοικητικά, επιμελητιακά, χρειαζόμαστε υπολογιστές. Μόνο και μόνο για να ενημερώσουμε, για να επιτρέψουμε να αντιληφθούν πώς γίνεται η δουλειά. Όταν εκπαιδεύουμε το γενικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, το προσωπικό του Γενικού Επιτελείου, χρειάζεται να δώσουμε στοιχεία σχετικά με την ε, ηγεσία, με την ηγετική στάση. Μιλούμε, όπως υπόθηκε ήδη, για βασικό εξοπλισμό. Άρβιλα, στολές, αντίσκηνα, υπνόσακους. Και ε, φορεαμούς για να μπορούν να αποθηκεύουν και εξοπλισμό όπως ε, υπόστεγα στα στρατόπεδα για να μπορούν να φυλάσσουν τον εξοπλισμό τους στα όπλα τους. Το στρατιωτικό νοσοκομείο επίσης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα. Ελλείψη υπάρχουν στον εξοπλισμό, το νοσοκομιακό αλλά και σε φάρμακα. Και αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε. Οι εκπαιδευόμενοι. Στόχος μας είναι ο στρατός, στρατιώτες δηλαδή, που προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτούς εκπαιδεύουμε. Η επικοινωνία μας και με την ε, ηγεσία, την πολιτική και τη ερωτική των ενόπλων δυνάμεων ε, αφορά όχι μόνο τις ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην περιοχή του Μοκαντήσου, αλλά και γενικότερα και την υποστήριξη για τη μετακίνηση των στρατιωτών αυτών πέραν του Μοκαντήσου από άλλες περιοχές της Σομαλίας, ώστε να μπορούν να φτάνουν στο στρατόπεδο στο οποίο παρέχουμε την εκπαίδευση στο Μοκαντήσου. Και όπως πήγε ο κύριος Σικλόντι, Έχουμε ξεκινήσει και τη βιομετρική καταχώρηση με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ώστε να μπορούμε να ε, εντοπίζουμε και να έχουμε ευχερέστερη αναγνώριση των ε, εκπαιδευομένων. Από εκεί και πέρα θα είναι αρμοδιότητα της ε, ίδιας Σομαλίας να συνεχίσει τη δουλειά και να αξιοποιήσει μέσω των ενόπλων δυνάμεων της τους στρατιώτες αυτούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πάντως, κάποια στιγμή θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες τους μαζί με την άμεσα. Ε, Νομίζω αυτά ήταν για μένα. Α, Ο κύριος Σικλόντι. Ε, όποτε θέλετε με τη σειρά. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση την οποία θέλω να απτύξω περισσότερο. Όπου υπάρχουν εθνοφυλακές είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται πολιτικές ε, της κυβέρνησης που να μπορούν να ενσωματώνουν τα μέλη αυτών των εθνοφυλακών στις δυνάμεις τους. Στο να τους ε, αφήνουν για πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, δηλαδή στο περι... Ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιθώριο δεν βοηθάει. Το αντίθετο. Άρα ο στόχος θα πρέπει να είναι όποιος είναι διατεθειμένος να ενταχθεί στην σωστή παράταξη, σωστή πλευρά και να εγκαταλείψει αυτές τις ένοπλες δυνάμεις, τις ένοπλες ομάδες, θα πρέπει να έχει αυτή την ευκαιρία. η κυβέρνηση Σομαλίας έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο μια πολιτική αμνίστευσης των λιποτακτών και αρκετοί μάλιστα και ηγετικά στελέχη της ε, Al-Shabaab παραδόθηκαν. Οι δύο βέβαια πιο σκληροί έμειναν και που ήταν, ε, δεν περιμέναμε ασφαλώς να εγκαταλείψουν τις οργανώσεις τους και να παραδοθούν. Αλλά είναι νομίζω πολύ σημαντική αυτή η πολιτική της αμνηστίας εν γέννη, να και μιλούμε για νοικοδόμηση κράτους. Είτε το θέμα μας είναι τα παιδιά που στρατολογούνται, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή του κράτους δικαίου στη χώρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τους ε, στηρίξουμε με τις συμβουλές μας για να φτιάξουν το κράτος δικαίου. Ένα παραδείγματι πέραν της ε, κατάρτισης και εξοπλισμού του UTM στη Σομαλία. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται γενικότερα. Στην κατάρτιση και θαλασσιών δυνάμεων χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό πλαίσιο και τη νομική βάση. του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ιδρυθεί ένα κράτος το οποίο σέβεται το κράτος δικαίου. Γιατί δεν θεωρείται αδίκημα η πειρατεία στη Σομαλία σήμερα. Αμαρτία μπορεί να θεωρηθεί, αλλά όχι ποινικό αδίκημα. Η ιδέα ατιμορρησία είναι ένα γενικό φαινόμενο, γενικευμένο και στη Σομαλία, αλλά και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, σε πολλές περιοχές. Άρα εδώ μιλούμε για νοικοδόμηση κρατικών δορμών και ακόμα και μικρά μικρά βήματα μέσω της κατάρτισης των τα κτλ. μπορούν να φέρουν κάποια αποτελέσματα εάν τα δούμε μέσα στη γενικότερη προσπάθεια για την οικοδόμηση του κράτους δικαίου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα μόλις δούμε να ρίχνονται τα θεμέλια τουλάχιστον αυτού του κράτους μέσω του κράτους δικαίου. Και κάτι ακόμη, Ελπίζοντα ότι δεν έχω λησμονήσει πολλέ από τι ερωτήσει. Η θετική πορεία της χώρας, ρώτησε ο κύριος Κούκαν. Ναι, πάλι σε σύγκριση με τη γύρω περιοχή. Έτσι, αν κοιτάξουμε το Ιράκ και τη Συρία, προφανώς είναι πολύ πιο ε, θετική η εικόνα. Πολλές προσπάθειες γίνονται. Στο γιο στους λήψους συζητούσαμε πριν από λίγο τη Λιβύη, που είναι και θέμα των ε, Υπουργών των Εξωτερικών σήμερα. Αλλά δεν υπάρχουν λιβικέ αρχέ. Υπάρχουν. υπάρχουν εκπρόσωποι τη κυβέρνηση Λιβύη με, με του οποίου δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Άρα δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Άρα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί με την Σομαλία η κατάσταση να μην είναι ρόδινη. Αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση, έστω ομοσπονδιακή, που δεν τη χάνει τη ε, υποστήριξη όλων των πλευρών απαραίτητα τη αναγνώριση, αλλά πάντως κάτι υπάρχει και εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από ότι εγώ την περιοχή βλέπουν την εξέλιξη και μου λένε ότι είναι πολύ καλύτερες οι προοπτικές. Άρα υπάρχουν θετικά, ενθαρρυντικά σημάδια. Ε, για μας πρόκληση είναι να εντοπίσουμε τα θετικά σημάδια, να τα ενισχύσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι κάνουμε είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και επίσης και εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, λέει ο στρατηγός Μάντζη, Από τα θετικά σημάδια. Συνήφθη μια ε, συμφωνία πρόσφατα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών. Συμφωνία που αφορά την ενσωμάτωση των εθνοφυλακών στις διάφορες, των διαφόρων περιοχών στον εθνικό στρατό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Το στρατηγό. Θεωρείτε ότι καλύψατε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ακούσουμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων από ό,τι βλέπω. Πάντως θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να αποφύγουν τις κατασυρωήν ερωτήσεις, γιατί δυσκολεύουν πολύ τους ε, ομιλητές μας. Πώς να απαντήσουν σε τόσες ερωτήσεις. Μη λένε για δημητριακά εδώ Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα και τμήμα της συνεδρίασης. Ευχαριστώ τον αντιστράτηγο Αντώνιο Μάτζη που μας ενημέρωσε. Καλό τον Διευθυντή Κλόντι να παραμείνει για να μας ενημερώσει για τις ε, συνθήκες που έχουν σε σχέση με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλαχού. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Could you please conclude your chats? Thank you. Να σταματήσουν οι συνομιλίες παρακαλώ για να περάσουμε στο σημείο 5 της Μέσιας Διάταξης. Παρακαλώ τον Διευθυντή Ικλόντι Διευθυντή Γκάμπορ Ικλόντη. Σας υπενθυμίζω τη Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού, CMPD. ο οποίος έχει το καθήκον τώρα να μας ενημερώσει για τις ε, αποστολές και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα εξή έχω να σας πω, επειδή δεν είναι και πολύ ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές σκέψεις για τις αποστολές και επιχειρήσεις. Δεν θα καλύψω και τις 16 επιχειρήσεις και αποστολές. Εκτενώς θα εστιάσω σε κάποιες από αυτές τις πιο ενδιαφέρουσες και στη συνέχεια θα, θα πω δύο λόγια και για τις ενδεχόμενες μελλοντικέ δεσμεύσεις μας. Τι μέλη γενέστε, τι προβλέπετε στο μέλλον. Εν είδη ε, αυτά και ανάλογα μετά με τα δικά σας ερωτήματα θα δούμε που θα μας πάει το ταξίδι στη, στο δεύτερο ημίση αυτής της συνάντησης. Λοιπόν, κάποιες γενικές σκέψεις καταρχάς, όπως γνωρίζετε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 12 ετή περίπου εμπειρία σε αποστόλες και επιχειρήσεις. Ε, η πρώτη το 2003, και το καιρό δηλαδή, συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 34 ε, αποστολές και επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το διάστημα. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και επί του παρόντος ε, τρέχουν 16 από και Και αυτό δείχνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αριθμών, 34 και 16. Άρα είχαμε τη δυνατότητα και να ξεκινήσουμε νέες ε, αποστολές, αλλά και να κλείσουμε ενδεχομένω ορισμένες από τις ε, αποστολές και επιχειρήσεις αυτές. Κάποιες φορές ε, είναι πιο δύσκολο να βρει κανείς την πόρτα της εξόδου παρά την πόρτα της εισόδου, άρα αυτό μπορεί να το θεωρεί κανείς επιτυχία. Δεύτερον, Δείχνει αυτό ότι το 16 είναι παρόλα αυτά ένα μεγάλο νούμερο, όπως είπα, ιδίω εάν το βάλουμε στο πλαίσιο και το συγκρίνουμε με τους πόρους που έχουμε διαθέσει για τη στήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων ΕΠΑ. Συνολικά, από τις 16 αποστολές και επιχειρήσεις, οι 5 είναι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι τρει έχουν εκτελεστική εντολή, δύο εκπαιδευτικέ στο Μάλι και ε, Σομαλία δεν έχουν. Και έχουμε και 11 μη στρατιωτικέ ε, αποστολέ. Συνολικά το προσωπικό που έχει αναπτυχθεί σε αυτές τι αποστολές ανέρχεται στις 7.000 κατά το ίμιση στρατιωτική και οι υπόλοιποι όχι από ε, από το προσωπικό αυτό οι 600 περίπου που έρχονται από χώρες εταίρους, ένα 8% δηλαδή. Και αυτό από τη μια είναι καλό, γιατί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη από την αρχή από το 2003 σχεδόν όλες οι αποστολές και επιχειρήσεις ήταν ανοιχτέ, μπορούσαν σε αυτές δηλαδή να συμμετέχουν ε, και χώρες εταίροι. Από την άλλη πλευρά, αν δείτε για παράδειγμα την πιο πρόσφατη αποστολή μας, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συγκεκριμένα συνολικά 60 άτομα ήταν η εγκεκριμένη σύνθεση, νομίζω. Ότι έγινε και μία διάσκεψη για να συγκροτηθεί αυτή η αποστολή. Τέλο πάντων δεν είναι τόσο ροδινικό, να θα σας τα πω πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Χρηματοδότηση σίγουρα είναι ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, οι μη στρατιωτικές αποστολές χρηματοδοτούνται μέσω του προπολογισμού της ε, ΚΑΠΑΠΑΑ. περιορισμένος ο προϋπολογισμός, 260 ε, εκατομμύρια ήταν ο περσινός προϋπολογισμός, δεν είναι και μεγάλο αυτό το ποσό τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο όχι στο επίπεδο ε, της Ένωσης. Οι στρατιωτικές αποστολές τώρα χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού Αθήνα, αλλά μόνο μέρος του κόστους χρηματοδοτείται γίνεται αποδεκτό ως κοινό κόστος και επομένως περνάμε σε αυτό το μηχανισμό. Και όπως βλέπετε στο υπόλοιπο ποσό, εδώ μιλάμε για το 10% μόνο του συνολικού κόστους. Ο πρόεδρος Ελεντιών στο Μιλάνο έλεγε ότι η αλληλεγγύη μας είναι 10%. Δεν κατάλαβε κανείς τι εννοούσε και το εξήγησε. Αν μόνο το 10% δηλαδή γίνεται αποδεκτό ως κοινό κόστος, μπορούμε έτσι να μετρήσουμε για την αλληλεγγύη. Άρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να είναι σαφές ότι το κόστος και ο προπολογισμό της δεν είναι πάντοτε τόσο χαμηλός. Ε, ε, είναι συνδετή απόφαση των κρατών μελών να παραμένει σε αυτά τα τόσο χαμηλά επίπεδα και όχι μόνο για μια χρονιά. Μιλάμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επτά χρόνια δηλαδή θα είναι έτσι κατάσταση. Άρα έχουμε δεμένα τα χέρια. Εδώ μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια τεράστια αντίθεση που θα διευρύνεται περισσότερο μεταξύ της φιλοδοξίας που έχουμε να υψώνουμε την, ευραϊκή, την ευρωπαϊκή σημαία οπουδήποτε υπάρχει κρίση. Και σε σχέση με τους πόρους που διαθέτουμε. Και όταν μιλάμε για πόρους, δεν μιλάμε μόνο για οικονομικούς πόρους, μιλάμε για τη συμβολή, τη συμμετοχή προσωπικού, σε αυτές τις αποστόλες και επιχειρήσεις. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Εύκολο θα ήταν να πω ότι αυτή είναι η πόρη που έχουμε στη διάθεσή μας, άρα θα πρέπει να κατεβάσουμε τις ε, φιλοδοξίες μας και μάλιστα σημαντικά. Είναι όμως αυτό κάτι που επιθυμούμε και που μπορούμε να το επιτρέψουμε για την Ένωση. Δεν νομίζω επομένω είναι σημαντικό δεδομένης ε, της ε, ακαμψίας ε, των οικονομικών χρηματοδοτικών κανονισμών και της ερμηνείας ορισμένων μέσων και εργαλείων να αρχίσουμε να αλλάζουμε νοοτροπίες και να ρίχνουμε τα τείχη που χωρίζουν τα διάφορα εργαλεία και μέσα, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ευελιξία. Και για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ένωσης. Πολύ συχνά το ίδιο πρόβλημα ισχύει και στα κράτη-μέλη. Εγώ έχω εργαστεί και ε, στη χώρα μου και έχω δει και αλλού και τις ίδιες ε, παραμέτρους να επηρεάζουν. Αναπτυξιακοί στόχοι που ε, με τους στόχους της ασφάλειας. Ε, μιλάμε για δύο διαφορετικά σύμπαντα, δύο διαφορετικούς κόσμους να μιλάμε για μια σφαιρική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να την ασκούμε όμως αυτή την προσέγγιση και σε εθνικό επίπεδο. Άρα πρέπει κάπως ε, καλύτερα και πληρέστερα να συντονίζονται τα συμφέροντα τα, των κρατών εσωτερικά. Δηλαδή, τα συμφέροντα τα εξωτερικ... της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας μιας χώρας είναι εντελώς διαφορετικά από τα συμφέροντα ή τις ε, ενέργειας μιας χώρας, της ίδιας χώρας στον τομέα της ε, ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξει μια μετακίνηση σε διεθνές επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένουμε πραγματικά κάποιες ρηξικέλευτες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. About financing. Uh, against fourth generation is a problem. Α, η δημιουργία ε, δυνάμεων, force generation. Είναι ένα ζήτημα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, U for RCA, είναι μοντέλο. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Μπορεί να δράσει τόσο γρήγορα η Ένωση. Αυτό δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε πάντοτε όλοι μας. Παραδείγματος χάρη όταν η U4 RCA ...79 μέρες μετά τη λήψη απόφασης χρειάστηκε ε, για να, περάσουν για την ανάπτυξη. 79 μέρες. Γιατί ήταν παράδεκτα μεγάλο το χρονικό διάστημα για τη χρήση μιας μάχημης ομάδας ήταν μια χρυσή ευκαιρία και χάθηκε εντελώ με εξωθρύντο τρόπο. Γιατί το battle group θα τέριαζε, γιατί έχει πολύ μεγάλη, μικρότερη προθεσμία, γύρω στις 10 μέρες. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε με τη φανταστική αυτή ιδέα των μάχημων ομάδων, τα battle groups. Χρειάστηκε ένα είδος γεφύρωσης μιας επιχείρησης γέφυρας. Το U4SEA ευρωπαϊκής πλευράς ήταν κάτι που θα ήθελα να χρησιμοποιήσουν λοιπόν ως μοντέλο και να το αναπαραγάγουν και στο μέλλον αν χρειαστεί. Ήδη ε, το να μιλάμε για γενικότερη ε, επανάληψη μήνυση αυτού του μοντέλου είναι κάτι ε, τραβηγμένο, ίσως υπερβολικό. Πάντως, αν ε, τα Ηνωμένα αργά κινούνται για την δημιουργία και ανάπτυξη δυνάμεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει και που έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Και μπορεί να παρασχεθεί και βοήθεια στον τομέα της διοικητικής μέρημνας κτλ. Άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που όμως κρύβει ένα ευρύτερο, το πρόβλημα της αλληλεγγύης. Αν λοιπόν μιλάμε για 60 άτομα που τα στέλνουμε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για να στηρίξουν έναν στόχο επί το οποίο συμφώνησαν ότι είναι σημαντικός και 28 χώρες μέλη. Αυτό βασίστηκε σε αίτημα του Πρόεδρου της χώρας. Και επειδή ο ΙΕ ξεκάθαρα είχε πει ότι δεν θέλει να παρέμβει πριν τις εκλογές στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Και πριν οριστεί νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρόβλημα αλληλεγγύης. και μία χώρα, η Γαλλία, δίνει το 60% αυτών των 60. Και κάποιοι από χώρες εταίρους που ενδιαφέρονται, όπως η Γεωργία για παράδειγμα, που πάρει προστασία. Η Μολδαβία έχουν στείλει επίσης άτομα. Το πρόβλημα όμως στο θεμείο δεν αλλάζει. Δεν θα μπορούσε η διάσκεψη αυτή για τη συγκρότηση δυνάμεων να προσελκύσει τα λίγα ουσιαστικά άτομα που χρειάζονταν για αυτή την αποστολή. Και συνήθως ε, αυτές οι αποστολές κοινής της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας προβλέπονται για μικρό χρονικό διάστημα, έχουν έναν στόχο συγκεκριμένο και αυτό περιορισμένο χρονικά και συνοδεύονται ως το δυνατόν από μια πιο σαφή στρατηγική αυτής εξ αρχής. Όμως, πολλά πρέπει να θυμόμαστε, μεταξύ των οποίων χρειάζεται στρατηγική εξόδου και είναι σημαντικό, αλλά καλό είναι να γίνει και σωστά είσοδος. γιατί το ένα εξαρτάται από το άλλο. Όπως είδατε ίσως, έχουμε πάψει να μιλάμε για στρατηγικές εξόδου και μιλάμε για μεταβατικές στρατηγικές, διότι από πολιτική πλευρά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι άπαξ και ληφθεί μια απόφαση. Η ανάπτυξη μια χώρα, η παροχή υποστήριξη στη χώρα αυτή, η Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Σομαλία ή οποιαδήποτε άλλη, Ουκρανία, Γεωργία, πείτε εσείς όποια χώρα θέλετε. Μιλάμε για μια μακροχρόνια δέσμευση. Η υποστήριξη μπορεί να δοθεί και με διαφορετικό τρόπο, αλλά θα πρέπει να δοθεί. Δεν συμβαίνει όπως τώρα με την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που είναι ουσιαστικά μια μεταβατική αποστολή. Έξι μήνες εμείς μετά μπαίνουν, ε, ε, μπαίνει ο ΙΑ και εμείς αποχωρούμε. Όχι, άπαξ και ληφθεί απόφαση πρόκειται για μια μακροχρόνια δέσμευση παροχής βοήθειας στην εκάστοτε χώρα. Και ξέρουμε ότι αυτό που θέλουν οι χώρες αυτές είναι η οικοδόμηση κράτους. Και αυτό σίγουρα δεν γίνεται μέσα σε έξι μήνες. Αλλά και στο μη στρατιωτικό σκέλος, δεν ξέρω αν το συστήσαμε, νομίζω, για την Ουκρανία ε, το είπαμε. Και τη μεταρρύθμιση του τομέα της πολιτικής ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει εντολική εντολή είναι για δύο χρόνια. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε δύο χρόνια ακόμη και σε μια φυσιολογική χώρα που δεν βρίσκεται σε τέτοια κρίση ο τομέας της ε, ασφάλειας μπορεί να μεταρρυθμιστεί μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια είναι αδύνατον. Είναι πάρα πολύ πιο μακροχρόνια αυτή η δέσμευση, ιδίω σε μια χώρα που δεν τα έχει καταφέρει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της ε, για μεταρρυθμίσεις κατά το παρελθόν τα τελευταία 20 χρόνια και που τώρα ένα μέρος της ε, ε, είναι κατεχόμενο και υπάρχει πόλεμος, άρα το επιχείρημά μου είναι Αυτές οι επιχειρήσεις σχεδόν χωρίς καμία εξαίρεση είναι μακροχρόνιες, μακρόπνες. Κλείσαμε κάποιες, είχαμε 34, είπαμε στις 16 ορισμένες δηλαδή τις ολοκληρώσαμε. Υπάρχουν και κάποια μεταβατικά στάδια σε κάποιες περιπτώσεις ε, όπως είναι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για παράδειγμα από το καλοκαίρι και μετά θα έχουμε ένα είδος μικροαποστολής στο πλαίσιο της σταδιακής ε, κατάργησης και στην Αταλάντη που μπορεί να μεταβούμε σε μια άλλη φάση, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Το Γιούλεξ, κοσυφοπεδιο μπορεί και εκεί να έχουμε μια μετάβαση, να περάσει ε, στις τοπικές αρχές κτλ. Ε, κτλ όλα αυτά πρέπει να τα καταγράψουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να προχωρήσουμε ιδανικά δίνοντας την εξουσία στις τοπικές αρχές. Αν όχι σε άλλους διεθνείς ε, φορείς, σε ένα άλλο, πιο μακρόπνο ευρωπαϊκό εργαλείο και μέσο. Όπως αυτά που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι αποστολές και δράσεις είναι ένα εργαλείο από την εργαλειοθήκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει κρίση κάπου στον κόσμο και μας ασκούνται πιέσεις να αντιδράσουμε κάποιο τρόπο. Η άμεση αντίδραση πρέπει να είναι αμέσως να αναπτύξουμε μια αποστολή. Γιατί αυτό μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση. Το καλύτερο μέσο. και δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται αυτές οι αποστολές της ε, κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας παρά μόνο εάν απαιτείται αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με αντίθετος φυσικά. Κάτι ακόμη, τελευταία παρατήρηση γενικού χαρακτήρα για να προχωρήσω και το έχω αναφέρει νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δυναμικού σε επίπεδο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό. Δηλαδή αποστολές κατάρτισης όπως αυτές τις οποίες παρουσίασε ο στρατηγός Μάτζη, Ουκρανία και άλλες προσπάθειες. Σε αυτό είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα είμαστε μια υπερβολικά μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να απτύξουμε επιχειρήσεις τύπου ΑΕΣΕΦ. Δεν ιδιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους δράσεις. Πρέπει να βρούμε τις ευκαιρίες μας αλλού. Ευκαιρίες υπάρχουν και ακριβώς στο τομέα της ανάπτυξης του δυναμικού υπάρχουν. ακριβώς την ανάπτυξη του δυναμικού που μπορεί να υπάρχει στο μέλλον. Στο Ιράκ και το ίσις, επαραδείγματι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο να καταπολεμήσει την, ε, το ΙΚΙΛ, ούτε καν προσπαθούμε διότι θα ήταν και επικίνδυνο να λάβουμε κάποια δράση ουσίας στη Λιβύη. Γιατί όμως να μην προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε χώρες της περιοχής όμορες με αυτό το πεδίο της κρίσης που δεν έχει επηρεάσει όμως ο ιός της, ε, του ΙΚΙΛ αφού υπάρχει τη δυνατότητα και έτσι να μπορέσουν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Είτε πρόκειται για την Ορδανία ή τον Λίβανο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες θα ήταν δεκτικές. Και άρα αντί να προσπαθούμε να αντιδρούμε στα προβλήματα ε, και να τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, ας προλάβουμε τις εξελίξεις. Να σταματήσω εδώ το θέμα αυτό για να περάσω σε κάποιες τρέχουσες επιχειρήσεις. Ξεκινώ με κάτι που θεωρώ όχι ως επιχείρηση αλλά πολύ επίκαιρο θέμα γιατί ήταν θέμα και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ε, αυτές τις μέρες Λιβύη. Σας ενδιαφέρει φαντάζομαι ιδιαίτερως και σας. Αν κοιτάξουμε λοιπόν την κατάσταση στη Λιβύη, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση σχετική με την ασφάλεια είναι ιδιαίτερα πτυτική και πάντως μη βελτιούμενη. τους επιδεινώνεται διαρκώς. Οι προοπτικές πολιτικού διαλόγου πολύ αβέβαιες. Προσπάθειες του Μπερνάρντι των Λεών, τεράστιες προσπάθειες, αλλά αποτελέσματα δεν έχουν φέρει, ορατά τουλάχιστον. Η δε πιθανότητα για μια γενική κατάπαυση, για μια γενική εκχειρία, ε, ώστε να επιτρέψει την ε, επιβίωση της, τη δημόρφωση μάλλον μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι πολύ χαμηλές. Εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας, η ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών που θα μας έδιναν ε, την εντολή να αναλάβουμε δράση. Πέραν των λοιπόν συνθήκων δεν βλέπετε να υπάρχει. Πιθανολόγηση της αποδοχής από τη Λιβύη ε, μιας τέτοιας αποστολής στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας επίσης δεν προβλέπεται. Είναι μάλλον απίθανο ή εντελώς απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή γιατί βέβαια μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση με λίγα λόγια έστω και υπεραπροστευμένα που αντιμετωπίζουμε. Με, όλες αυτές τις, ε, με όλα αυτά τα αβέβαια λοιπόν στοιχεία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις αβεβαιότητες, έχουμε μπορέσει να ετοιμάσουμε κάποια σχέδια για το μέλλον για να προετοιμαζόμαστε. Όταν έρθει η ώρα δηλαδή να αναλάβουμε δράση, να προσφέρουμε υποστήριξη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Και έχουμε κάποιους άρθρους στο μανίκι, με τη μορφή σχεδίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, βέβαια με την ε, προϋπόθεση θετικών εξελίξεων στον διάλογο, την ε, πρόβλεψη πώς θα μας ζητήσουν συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένη υποστήριξη αρχές της Λιβύης λοιπά. Όλα αυτά αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για τον σχεδιασμό μας, γιατί ο σχεδιασμός γίνεται εν κενό εκεί που χρειαζόμαστε δηλαδή να σχεδιάσουμε κρίσιμες υποδομές, είτε πρόκειται για λιμάνι, είτε πρόκειται για αεροδρόμιο, άλλες υποδομές, ποιος θα αποφασίσει τι είναι αυτό που χρειάζεται. Άρα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που συζητούμε είναι μια ευρέως, ε, με ευραία υποστήριξη πολιτική προσέγγιση για τη Λιβύη και μια ευέλικτη ανταπόκριση βέβαια στο πεδίο της ε, ε κοινή πολιτικής άμυνας γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Άρα η κατάσταση μένει έτσι. Και όπως είπα, ο σχεδιασμός είναι εν κενό ουσιαστικά. Τι μπορούμε να κάνουμε εάν και εφόσον προκύψουν οι δυνατότητες. Και αυτό υπό τον όρο ότι και οι Λίβοι συνομιλητές μας θα ζητήσουν την υποστήριξη, εάν σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και διατυπώσει ένα συγκεκριμένο αίτημα για επέμβαση και υποστήριξη στα Ηνωμένα Έθνη ή ψήφισμα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που να εξασφαλίζει εντολή για μια αποστολή δική μας. Αυτά όλα βέβαια μένουν ε, στο χώρο των ευσεβών πόθων Και αυτό που γίνεται, ή τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να πράξουμε, είναι να αναπτύξουμε μια προσέγγιση σε δύο φάσεις. Πρώτα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με την κατάσταση που έχουμε. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε στο μια μικρή ομάδα επιχείρηση για να υποστηρίξουμε την UNSMIL στην, ε, με σχεδιασμό των ΗΠΑ γιατί έχουν περιορισμένες δυνατότητες σχεδιασμού και έτσι ταυτόχρονα έχουμε και εμείς μια ματιά στο πώς λειτουργεί ε, η UNSMIL και προς τα που πηγαίνει η κατάσταση. Χρήσιμο πάντα. Αυτό όμως μόνο μια μικρή αποστολή. Όλοι οι άλλοι φίστανται τα πειρά και περιμένουν να βελτιωθεί η κατάσταση. Και κάποια πρόσθετα σχόλια όταν έρθει η ώρα. Θα είναι κέρια σημασία οι αρχές της Λιβύης να εκφράσουν ύψες του επίπεδου στράτευση και προσήλωση, αλλά ταυτόχρονα και η περιφερειακή εταίρη, τα άλλα κράτη, για ό,τι είναι να γίνει, για ό,τι δράση να αναλυφθεί. Και βεβαίως θα χρειαστεί και εμείς να έχουμε μια σαφή, σαφώς σχεδιασμένη στρατηγική. Για δύο λόγους τουλάχιστον, καταρχάς για την επιτυχία της ε, ε, αποστολής, που είναι πάντα ένα πρόβλημα, αλλά δεύτερον και για να ε, ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες, γιατί ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει αυτή η δουλειά, όταν ξεκινάει μια επιχείρηση, οι προσδοκίες είναι υψηλές και πρέπει πάντα να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Η υποστήριξη των δυνάμεων. Η προστασία των δυνάμεων είναι πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το λέω αυτό διότι η Λιβύοι δεν είναι ούτε και πρόκειται να γίνει ακόμη και αν σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ε, ενότητας, ακόμη και αν μας προσκαλέσουν, ακόμη και αν αναλάβουν και τα Ηνωμένα Έθνη το ρόλο και μας δώσουν εντολή, δεν πρόκειται να καταστεί η Λιβύη περιβάλλον πρόσφορο. Γιατί είναι πολλές τρομοκρατικές δυνάμεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και είναι σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ή και βούληση για εξασφάλιση προστασίας των δυνάμεων. Άρα είτε μένουμε στα χέρια της, ε, των αρχών της Λιβύης, είτε πρέπει να διαμορφώσουμε την εμπλοκή μας κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να τη διαχειριστούμε, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο. Για τη Λιβύη νομίζω αυτά έχω να πω. Για τη Σομαλία μιλήσαμε. Καλύφθηκα επομένως. Η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, έχουμε σχέδια για αποστολές τον Ιούλιο στο Σουδάν και μετά στις, ε, ε, στα κεντρικά της Αταλάντα το Σεπτέμβριο που θα επισκεφθούμε τη Βοσνία Ερσεγοβίνη αργότερα. Ίσως θα είναι σκόπιμο λοιπόν, αν και πάντα θα έχουμε δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε πριν από τα ταξίδια μας. Θα ήταν όμως σκόπιμο να μας δώσετε και εσείς μια ε, επισκόπηση της εικόνας και πιθανά προβλήματα που μπορείτε να εντοπίσετε. Ίσως και συνάδελφοι να έχουμε άλλες ερωτήσεις. Μολδαβία. Ναι. Μάλιστα, στη Μολδαβία δεν έχουμε αποστολή ακόμα. παρόλα αυτά. Για τη Βοσνία και την Αταλάντη, αυτά ήταν τα τρία θέματα. Α, όχι, ας πω κάτι για τη Μολδαβία, λοιπόν. Δραστηριοποιηθήκαμε στην Ουκρανία και αν θέλουμε να βρούμε σωστές απαντήσεις για την ανταμετώπιση της κατάστασης στην Ουκρανία, τότε πρέπει να προσέξουμε και τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Τουλάχιστον να τις βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν το καινούργιο, τις καινούργιου είδους μικτές απειλές. Κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό. Η Μολδαβία, η Περθενιστερία, εκεί γίνονται κάθε μέρα προβοκάτσιες. Και περιμένουμε τη στιγμή να αντιδράσει η ηγεσία των χωρών αυτών. Όπως η φόλα που ρίχνουμε στη μέση και περιμένουμε να ορμήξει κάποιος. Να τις βοηθήσουμε λοιπόν, αυτό δεν απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, αλλά οικοδόμηση δυνατοτήτων. Ας πούμε το πολύ καλό πρόγραμμα Twinning της Επιτροπής ε, διδημοποίησης, δηλαδή αποστολής ειδικών από τα διάφορα υπουργεία για να βοηθήσουν για θέματα ασφαλείας διαδικτύου, τέτοια πράγματα που θα τους άρεσαν πολύ το ζήτησαν ήδη, μπορούμε να το χορηγήσουμε και άρα γιατί όχι. Τώρα με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας είναι βέβαια εκτός από, τις, από το πεδίο της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά πρέπει να βοηθηθούν και γι' αυτό οι χώρες αυτές. Ας πούμε ένα συμβουλευτικό ρόλο. Πώς να, πώς να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη που χάθηκε στην ψυχή των Ουκρανών προς τους διεθνούς οργανισμούς. Πώς να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό μια δημοκρατική αστυνομία με λογοδοσία, εθνοφυλακή κτλ. Και αυτά, και αυτά, και αυτά. Να ενδυναμωθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας σε τέτοιου είδους υβριδικές απειλές ή στρατηγική επικοινωνία προβλήματα δηλαδή και μέσα και έξω. Και μέσα και έξω. Αυτό για τη Μολδαβία. Τώρα θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η Μολδαβία είναι μικρή χώρα, ίσως η πτωχότερη της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί και αυτή να συμβάλλει στις αποστολές μας ας πούμε. Έστειλαν έναν στο RCA, Συγκέντρωση Αφρικανική Δημοκρατία δηλαδή. Παρά το ότι είχαν μόνο έναν να στείλουν, τον έστειλαν. Αυτά είναι μικρά βήματα, αλλά δείχνουν τη θέληση μιας χώρας να συμμετάσχει και να συμβάλλει. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος για το θέμα της ασφαλείας και άμυνας έχει περάσει πάνω από μισό χρόνο που από τότε που οι σχέσεις Ένωσης και Ουκρανίας, Γεωργίας, Μολδαβίας βελτιώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο με την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ένωση. Σήμερα τι προσφέρει η Ένωση στις χώρες αυτές αφού υπογράφτηκαν αυτές οι συμφωνίες για να ασφάλεια και άμυνα λέω. Τι περισσότερο προσφέρει τώρα από ό,τι πριν 2, 3, 4 χρόνια. Η απάντηση είναι μηδέν. Και πρέπει αυτό να αλλάξει, πρέπει αλλάξει. Για την Αταλάντη. πολύ επιτυχής ε, επιχείρηση σίγουρα. Ε, εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν επαναληφθεί πειρατικές απειλές. Το πρόβλημα είναι πώς να πιστούν οι χώρες μέλη, οι κυβερνήσεις να διατηρήσουν μια επιχείρηση ζωντανή εφόσον δεν υπάρχει πια το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα δεν εκμηδενίστηκε το φαινόμενο της πειρατείας στη θάλασσα έχει προς στιγμήν εξαφανιστεί, αλλά άμα φύγουν τα πλοία αυτά θα ξαναέρθει η πειρατεία. Πώς να πείσουμε λοιπόν τις κυβερνήσεις ότι το να κρατήσουμε δύο-τρία πλοία της Αταλάντης είναι καλή επένδυση. Πώς να διασφαλίσουμε ότι εκτός από την πειρατεία η Ανταλάντη θα μπορούσε να λύσει και άλλα προβλήματα και να αναλάβει και άλλες ευθύνες και άλλες στην Ανταλάντη υπάρχουν τουλάχιστον τρία στοιχεία που πρέπει να κρατηθούν πέραν της πειρατείας. Ένα είναι... Α? Ε? ένα είναι λέγω ότι έχει καθοριστεί και από τις χώρες μέλη και στις χώρες εταίρους αλλά και από τις βιομηχανίες ότι πρέπει να προστατεύονται να προστατεύεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πώς να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι η πληροφόρηση η... θα διατηρηθεί και η διανομή των πληροφοριών σε τόσο σημαντική περιοχή για μας. Δεύτερον, το γάμα 2. Η Αταλάντη έχει κινητοποιήσει, μπορεί να κινητοποιήσει πλοία υπό ενωσιακή σημαία για να κάνουν ορισμένες αποστολές. Αποστολάς. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Μιλήσαμε για την Ιεμένη πριν, Πριν από μερικές μέρες ή τις προάλλες ακούστηκε η ιδέα ότι η Αταλάντη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του τεράστιας ροής προσφύγων από την Ιεμένη προς τη Σομαλία. 260.000 ή 500.000 άνθρωποι. Τεράστιο κύμα. Λοιπόν, Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την Αταλάντη για να τους βοηθήσει συνοδεύοντας και προστατεύοντας τους. Την περασμένη εβδομάδα η Αταλάντη είχε τέσσερα πλοία που συνόδευαν 55 άλλα πλοία εξών 20 με νοσιακή σημαία. Δεν ήταν μόνο η Αταλάντη λοιπόν, αλλά κι άλλα, και άλλα πλοία, κι άλλα. Το γάμα 2 λοιπόν, άμα διατηρηθεί, μπορεί να κινητοποιήσει καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τυρόπο. Τρίτον, να μπορέσουν να αν οικοδομηθούν δυνάμεις γρήγορα. Αν υπάρχει μια κατάσταση ας πούμε που αποτεί άμεση ανταπόκριση, αντί να αρχίσουμε από την αρχή να σκεφτόμαστε τι λύσεις να εφαρμόσουμε, η λύση υπάρχει. Απλώ πρέπει να αναδημιουργηθεί η δύναμη. Πώς να τη συνδέσουμε με με την θαλάσσια στρατηγική, το ασχέδιο δράση για τη θαλάσσια στρατηγική που ενέκρινε πρόσφατα η Ένωση. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το κέρας της Αφρικής είναι περιοχή σημαντική για την Ένωση για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Ας πούμε η μεταφορά των αγαθών Θα δούμε πώς θα μπορέσει να μετατραπεί η Αταλάντη σε κάτι άλλο. Επίσης, τι κάνουν οι άλλοι παράγοντες όπως το ΝΑΤΟ. Έχουμε την επιχείρηση Ocean Shield αλλά τώρα δεν έχει εκεί κανένα πλοίο. Και η εντολή της Ocean Shield λύγει και αυτή. Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση με πρώτο τον κύριο Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση. Μας δείξατε πού δραστηριοποιούμαστε, πού υπάρχουν ελλείψεις, πού δεν ε, έχουν τόσο πολύ κίνητρο τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν και αν ε, δεν απατώμε, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή όχι. Άρα κάποια προθυμία υπάρχει. Σταχυολογώντας κάποια θέματα αυτό ο διαβόητος μηχανισμός Αθηνά. Νομίζω επιγόντως πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Δεν έχω καταλήψει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μετατραπεί σε κάτι άλλο δεδομένης της πραγματικότητας, ότι δηλαδή πολλές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Και αν ε, συνεχίσει, όσοι έχει βέβαια, ε, ενώ απαιτεί από άλλα κράτη να κάνουν πιο συχνά πράγματα ενώ έχουν ήδη υπερφορτωθεί με υποχρεώσεις. Γι' αυτό και περιμένω να έχουμε και σαφώς, σαφείς εναλλακτικέ εγγράφους. Νομίζω θα έχουμε πριν από την διάσκεψη κορυφής το έγγραφο αυτό, γιατί πρέπει να μεταρρυθμιστεί αυτός ο μηχανισμός, κατεπηγόντως. Σε τι αφορά το δικό σας ε, το ευθυνών. Ο σχεδιασμός ε, των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και οι δυνατότητες αυτές, πώς μπορούν να σχεδιαστούν από κοινού, τι μέτρα λαμβάνονται, τι πρόοδος έχει υπάρξει, μπορούμε να περιμένουμε κάτι ε, στις προσεχείς ε, εκδηλώσεις. Γιατί τη Λιβύη είπατε πολλά να αναγνωρίζουμε μια κάποια δομή στη Λιβύη, υπάρχουν ίσως και σε άλλες περιοχές. αλλά δύσκολα μπορούμε να έρθουμε σε κάποια βιώσιμη λύση. Τώρα, προστασία δυνάμεων. Αυτές οι μάχημες ομάδες, τα battle groups, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Θα ήταν ένα κατάλληλο εργαλείο για την προστασία των δυνάμεων. Να είναι πιο ασφαλή τα στρατηγία, η χώροι εκπαίδευση. Λόγω του μηχανισμού ε, εκπαιδευτικής εναλλαγής, κάποια στιγμή το πρέπει να γίνει και αυτό. Μπορούμε να εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Και άλλα σχόλια και ερωτήσεις θα είχα αλλά θα σταματήσω να δώσω το λόγο σε άλλους. Ευχαριστώ λοιπόν, κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και τη σχετική ειλικρίνεια στι επικρίσεις που απευθύνονται στα κράτη-μέλη. Φαντάζομαι ότι τι χρειάζονται. Πρέπει να τους καταγγείλουμε ισχυρίζονται ότι έχουν μια κοινή πολιτική ασφάλειας και αλλά μόνο το, κατ' όνομα είναι κοινή πολιτική. Και όμως έχουμε αρκετά θετικές εμπειρίες. Και ακούσα με χαρά και πάλι περιπτώσει όπου μπορέσαμε να αλλάξουμε κάτι ουσιαστικό όπως με την αποστολή Αταλάντη στη Σομαλία, αλλά και άλλες αποστολές, στρατιωτικές και μη. Όμως, αισθάνομαι μεγάλη δυσφορία και απογοήτευση ότι τα όταν βλέπω ότι τα κράτη-μέλη πώς δεν μπορούσαν και την εσωτερική κρίση να αντιμετωπίσουν, είναι αδύναμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και της ξένης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και γελάνε τους πολίτες. Αρκεί να κοιτάξουν όμως τη Μεσόγειο για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι δεν υπάρχει και πά. Εκεί που είναι πιο κοντά το πρόβλημα στις ακτές μας, στη Μεσόγειο. Κάθε μέρα θα βλέπουμε τις τις αυτές σκηνές των ανθρώπων που πεθαίνουν και πνίγονται στη Μεσόγειο. Κάθε άνοιξη η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότητα. Κάθε χρονιά γίνονται οι συγκρούσεις όλο και πιο βίες. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ευθύνες και εκπαραλήψεως, όπως συνέβη στη Συρία. Σε αυτό δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλεία με τον τρόπο λειτουργία του και η απουσία διεθνών συνθήκων. Για τη Λιβύη ιδέα που γνωρίζω πολύ καλά, ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε συνελθώ στο Κοινοβούλιο, γιατί την επισκέπτομαι τακτικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται όχι εκ της δράσεως, με την παρέμβαση κάποιων κρατών μας στη Λιβύη για να βοηθήσει τους πολίτες να ξεφορτωθούν το καντάφι, ο οποίος ήθελε να σφαγιάσει τους πολίτες του. Αλλά λόγω της αδράνειας στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσύ μόλι μόλις μας είπατε ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο το ζήτημα της αποστολής μιας αποστολής ε, ΚΠΑ στη Λιβύη. Τώρα που είναι άντρο τόσων τρομοκρατικών οργανώσεων η Λιβύη, όπως το ξέραμε πολύ καλά εξ ότι θα συνέβαινε, όπως πολλές φορές το έχουμε γράψει σε διάφορες εκθέσεις. Λυπούμε που δεν έφερα χειροορβομβίδα από αυτές που βρίσκει κανείς στο δρόμο εκεί. Ήταν τόσο εύκολο. Δεν μπορούσα να την είχα βάλει πάνω στο γραφείο κάποιου. Τώρα λοιπόν που αναζητούν ασφαλή λιμένα όλοι αυτοί οι απελπισμένοι στις ακτές μας, πάλι δεν κάνουμε τίποτε και όταν υπήρχε η περίοδος, η εποχή στην οποία μας παρακαλούσαν ο Πρωθυπουργό της Λιβύης, είχε έρθει και εδώ και στο ΝΑΤΟ και εκλυπαρούσε να αναπτυχθεί αποστολή. Πραγματικό πρόβλημα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι το αξεπέραστο εκείνη την εποχή, το ανυπέρβλητο ως πρόβλημα. Τώρα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση και συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Με όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Μπέναντι και τον επενούμε γι' αυτό. Αλλά χρειάζεται αποστολή ΚΠΑ στη Μεσόγειο με τι άλλο. Μάλλον δεν μπορούμε να στείλουμε στρατιώτες, ούτε καν ομάδες ε, μαχητικές battle groups που τους έως ποτέ δεν αναπτύχθηκαν. Αλλά εν αέρια και θαλάσσια αποστολή ΚΠΑ θα ήταν δυνατόν να αναπτύχθηκε και όφιλε να βρίσκεται ήδη στα νερά και τους εθέρες Λιβύης. Το ότι πνίγηκαν περίπου χίλιοι άνθρωποι προχτές στην ε, Μεσόγειο οφείλεται στο γεγονός ότι πήγε ένα πορτογαλικό αλλιευτικό σκάφος να βοηθήσει να προσφέρει αρρωγή στους ανθρώπους αυτούς που είχαν στείλει και πάνω στην αναστάτωση του ποιος θα βγει πρώτος ε, να περάσει στο πορτογαλικό σκάφος ανετράπει το αλληλευτικό των μεταναστών και έτσι πνιγήκαν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια επιχείρηση και πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι πιο σημαντικό, πιο ευρεία κλίμακος από αυτό που έχει γίνει στη Λιβύη όταν έρθει η ώρα και αν έρθει η ώρα για εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από αυτά που παρατηρήσατε για το οικονομικό, για την απουσία πόρων οικονομικών, δημιουργία δυνάμεων, Αποσία βούλησης. Ναι, αλληλεγγύη χρειάζεται. Σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα είναι η απουσία αλληλεγγύης. Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν και κράτη-μέλη τα οποία ξεκάθαρα μποϊκοτάρουν και υπάρχει ανάγκη, πέραν να επικρίνουμε όλα τα κράτη-μέλη, υπάρχουν κράτη τα οποία παρεμποδίζουν την ανάληψη ιασδήποτε αποφάσεως στο πλαίσιο είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ΝΑΤΟ. Ένα από αυτά είναι η Βρετανία. Με τα μου το λέω. Είναι υπεύθυνη και για την αδράνεια στη Λιβύη, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει μποϊκοτάρει την ΚΕΠΑ, τις δράσεις στην άμυνα, στη Λιβύη, σε ένα χώρο. Σας παρακαλώ να τελειώνετε κυρία μου, σας παρακαλώ, δεν έχω πολύ χρόνο. που λέει. Παρακαλώ. Ja chciałem zapytać przede wszystkim o misję EUBAN w Mołdawii i Ukrainie. Jej mandat po 10 latach... No... Για τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Πρόκειται να εκπνεύσει η εντόλη στερα από 10 χρόνια φέτος. Χρειάζεται όμως ακόμη περισσότερο από ό,τι ποτέ. από αυτά που μας είπατε. Εγώ καταλήγω στις σπέσμα ότι δεν πρέπει να λήξει. Πρέπει να παραταθεί μάλλον. Sorry. No. Uh, Mrs. Ceballos. Eh, då kan ni hålla lurarna på. jag fick svar på många av de frågor jag ställde redan. Men eh, ni talade om eh, Μιλήσατε για στρατηγική εξόδου και για μια διαφορετική στρατηγική που δεν θυμάμαι πια. Αλλά πάντως για μακροχρόνια δέσμευση. Εγώ όταν ακούω στρατηγική εξόδου σκέφτομαι και τι θα γίνει μετά την έξοδο. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχουμε στρατηγική εξόδου για τη Λιβύη αλλά πλήρες χάος. Όταν κανείς αναλαμβάνει μακροχρόνια δέσμευση, μπορεί ένα τμήμα να το αφιερώσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ένα άλλο τμήμα σε πολιτικές δραστηριότητες. Και αυτές οι πολιτικές δραστηριότητες μπορεί να αλλάξουν μέσα στο χρόνο, στην αρχή να χρειάζονται μερικά πράγματα και μετά άλλα και ύστερα πάλι άλλα. Είναι λοιπόν σημαντικό η, η μακροχρόνια αυτή δέσμευση να ακολουθεί μια λυσίδα ώστε να μπορεί κανείς τελικά να εμπιστευτεί όλες τις επιχειρήσεις στις τοπικές αρχές. Επίσης μιλήσατε για το Λίβανο και την Ιορδανία και για προληπτικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν εκεί. Σήμερα το Ισλαμικό κράτος είναι στα πρόθυρα εκεί. Τι προβλέπετε λοιπόν για υποβοήθηση αυτών των χωρών για πρόληψη. Υπάρχει τίποτε παραπάνω από την απλή στήριξη των στρατοπέδων προσφύγων. Έχει προβλεφθεί τίποτε άλλο για πραγματική βοήθεια του Λιβάνου και της Ιορδανίας για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση, κύριος Πρώην. Ευχαριστώ. Ένα πράγμα θέλω να πω στον, στην γείτονα και φίλη μου Άννα Γκόμες που μίλησε για τη χειροβομβίδα που κόντεψε να φέρει μαζί της από τη Λιβύη ούτως ή άλλως κάνει τόσο εκρηκτικά σχόλια που μια χειροβομβίδα δεν θα τις χρειαζόταν. Όχι εσύ Άννα, όχι, οποιοδήποτε άλλος, αλλά εσύ όχι. Ας παραμείνω όμως στη Λιβύη. Ήταν χώρα υποδικτατορία για πόσο 30 χρόνια παραπάνω και από ό,τι θυμάμαι πριν από τη δικτατορία ο βασιλεύς δεν ήταν επίσης κανένας μεγάλος δημοκράτης. Έχουμε λοιπόν δει τουλάχιστον δύο γενιές αντιδημοκρατικής πολιτικής και η ανησυχία μου για αυτή την αργή, τόσο αργή πρόοδο στη δημιουργία ικανοτήτων εξηγείται μεν, κυρίως από το ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί τι είναι οικοδόμησης έθνους. Watch them to... Θα περιοριστούμε λοιπόν να βλέπουμε αν θα κάνουν αυτό που θέλουμε να κάνουν, δηλαδή να δημιουργήσουν μια δημοκρατική διακυβέρνηση ή υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να τους βοηθήσουμε να το πράξουν όχι στρατιωτικά, αλλά στέλνοντας ανθρώπους που γνωρίζουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το άκουσα, ίσως εσείς ξέρετε κάτι. Γιατί έτσι θα κινούνταν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας να ζητήσω, να ρωτήσω και εγώ κάτι για τη γεωργία. Ιδίως για την αποστολή μετά την πιθανότητα να ληφθούν και άλλα ρωσικά μέτρα για την Οσετία κλπ. Επίσης, θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Σιλπερνιό μια προηγούμενη φορά για το πώς βλέπει ο κόσμος στην κεντροαφρικανική δημοκρατία τις ενωσιακές επιχειρήσεις και ορισμένες αμφιβολίες του. Γνωρίζουμε ότι είναι θετική η άποψη του κόσμου, αλλά παρόλα αυτά η ενδιάμεση γεφυρωτική αποστολή ήταν τόσο εξαιρετική που γενικά η αντίληψη του κόσμου, αλλά όχι μόνο του κόσμου, αλλά και των κυβερνητικών εκεί που Ρωσόπων, δείχνει ότι φοβούνται ότι όταν λήξει η αποστολή θα φύγουν οι εκπρόσωποι της. Ε, άρα πρέπει από τη μία να τους πείσουμε ότι έχουμε μακροχρόνια δέσμευση αλλά και από την άλλη ότι πρέπει να διαχειριστούμε και τις προσδοκίες να εξισορροπήσουμε αυτά τα δύο πράγματα διότι σίγουρα χρειάζεται Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά, έχετε και τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας είμαι ευγνώμων για το συνεχές ενδιαφέρον που δείχνετε. Το εκτιμώ όλος ιδιαίτερος. Yeah, uh, decisions are taken. Ναι, πράγματι λαμβάνονται με ομοφωνία οι αποφάσεις, δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υποστηρίζουν μια αποστολή για να λάβει χώρα. για τη χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες πληρώνουν, οι υπόλοιποι κάθονται και περιμένουν. Είναι μεγάλο το δίλημα. Τη μια πλευρά θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος να μετρήσει κανείς την αλληλεγγύη. Όλοι θα έπρεπε να συνεισφέρουν κανονικά, είναι μια κοινή απόφαση, άρα και 28 ως ομάδα αποφασίζουν την ανάπτυξη δυνάμεων, την άλυψη δράση σε ένα θέατρο επιχειρήσεων. Άρα θα έπρεπε να αναλάβουν από εκείνη την ευθύνη. Αν όμω ε, υπάρξει τέτοιο κανόνα προκύπτει μετά το ερώτημα κατά πόσον είναι εύκολο μετά να υπάρχει συνένεση, να υπάρχει ομοφωνία. Αν κάποιος δεν συμβάλλει και απλά αφήνει τους άλλους, ε, πιο εύκολα συμμετέχει, συνενεί όταν όμως πρέπει να χρηματοδοτήσει και υπάρχουν και άλλες συνέπειες, ίσως ε, μετριαστεί η προθυμία και των 28 να στηρίξουν μια επιχείρηση. Είναι ένα δίλημα λοιπόν. Ποια θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη λύση που από τη μια θα ενισχύει την ενότητα και την αλληλεγγύη των 28, κάτι που είναι πολύ αναγκαίο, θα βοηθά τον επερισμό των βαρών, χωρίς να απομίζεται το βάρος μόνο ένα κράτος, γιατί σήμερα φαντάζομαι ότι συζητάτε και την ανάπτυξη των μάχημων ομάδων, τα battle groups, αλλά και εδώ έχουμε αυτό το θεμελιώδες συζήτημα. Δηλαδή, γιατί Πράγματι, τεχνικά συμφέροντα παίζουν ρόλο. Άλλα συμφέροντα έχει η χώρα που ηγείται ενό battle group και είναι σε stand-by και άλλα μια χώρα που αποφασίζει να συμμετέχει σε ένα θέατρο, να σε ένα θέατρο επιχειρήσεων. Το είδαμε με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που κατά 120% ταιριάζει ε, στην περιγραφή ε, της χρήσης ενός battle group που δεν χρησιμοποιήθηκε όμως τελικά. Η Ελλάδα αναφέρεται επίσης συχνά ήταν σε stand-by το 2014 στο πρώτο εξάμεινο για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά δεν, υπήρξαν, δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Πέρα από δύο εβδομάδες είχαμε ένα άλλο, πέρα δύο μήνες, με το Ενωμένο Βασίλειο που έδειξε ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν εξαρτάται από το μέγεθος της χώρας και ακόμη και αν δεν, ε, εύκολα, δεν προσδίζονται εύκολα κάποια συμφέροντα, δηλαδή ποια χώρα θα αναπτύξει δυνάμεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καμία δεν θα έχει πολυζωτικά ζητήματα και ε, διακυβέρνοντα το με τη ασφάλεια. Αλλά σήμερα το ότι μπορώ να αναμένω, η αρχή ότι αναμένω αλληλεγγύη μόνο από εσένα, εάν εγώ δείξω αλληλεγγύη προ εσένα, θα έπρεπε νομίζω να, είναι λίγο, να λειτουργεί λίγο καλύτερα και ομαλότερα ως αρχή. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο δίλημα. Στατιωτικό και μη στρατιωτικό σχεδιασμό από εκείνου. Ότι αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό σίγουρα εμεί κάνουμε αυτό το σχεδιασμό, όχι όμω και την διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι θα έχουμε σε δύο χρόνια μια αναφέρωση του ΙΕΣ. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις δομές διαχείρισης κρίσεων που θα πρέπει να εξοθολογιστούν για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να καταργηθούν οι πιθανές αλληλεπικαλύψεις, αλλά ακόμη δεν γνωρίζω τι θα προκύψει από τη διαδικασία αυτή. Πάντως θα με επηρεάσει σίγουρα και εμένα προσωπικά η αλλαγή, άρα είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει το στομότερο δυνατό. Γιατί δεν είναι και μια διαδικασία που αρέσει σε κανέναν να την ε, επιμηκύνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προστασία δυνάμεων, ανάπτυξη battle groups. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα battle groups δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί στην πλήρη του σύνθεση, ίσως κάποια στοιχεία του. Ίσως ε, το κομμάτι της επιτήρησης αναγνώρισης ε, και πληροφοριών, ISR. Όταν είναι όριμες οι συνθήκες, είναι μια πιο σοβαρή εμπλοκή. Τα battle groups πράγματι όμως, ναι, και το ακούσαμε και δημοσία από τη Σουηδία για παράδειγμα, που είναι ο δικός της μισός χρόνος για τα battle groups και πριν και μετά τις εκλογές επιβεβαίωσαν οι Σουηδοί ότι είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν battle group αν χρειαστεί. Και αυτό θα πρέπει να το ακούμε και από άλλα κράτη-μέλη, ώστε να τον περισσότερο. Δηλαδή, αν υπάρξει δυνατότητα και μπορεί να αναπτυχθεί ένα battle group, έστω μια φορά. Καλό θα ήταν να δούμε πώς δρούν αυτές οι ομάδες. Οι στατιωτικοί αξιωματικοί βέβαια από την άλλη τελειοποιούν όλο και περισσότερο αυτή την ε, έννοια. Είναι όμως όλο και πιο ε, ρευστά τα πράγματα και ίσως προκύψει και μεγαλύτερη απογοήτευση. Γιατί το φάσμα των επιλογών ε, για τα battle groups θα είναι ακόμα ευρύτερο. Αν εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται λοιπόν, αυτό θα οδηγήσει σε απογοήτευση. για τη Λιβύη ναυτική επιχείρηση. Πολλά παίζονται θεωρητικά και πολλές είναι επιλογές. Και εξετάζονται διάφορες ε, εναλλακτικές. Τώρα αν θα ήταν η καλύτερη επιλογή μια ναυτική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της μαζικής εισρωής ε, προσφύγων και αποφυγή πνιγμών ή ε, τι να πω, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Πρώτα απ' όλα και κυρίως γιατί πιστεύω ότι πρέπει να στραφούμε κατά των διακινητών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γνωρίζουμε ότι το 80% των προσφύγων που προσπαθούν να φύγουν από τη Λιβύη και να έρθουν στην Ιταλία, την Ισπανία ή τέλος πάντων να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη συνοστίζονται στο Αγκαντές. Να παρακαλέσω λέει πρόεδρος να μην αναλωθούμε σε συζητήσεις τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και καλό θα ήταν να ακούσουμε απαντήσεις. Μάλιστα, ναι, πράγματι είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό που θα απαιτήσει πολύ συντονισμό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, Interpol, Frontex, υπάρχουν όλοι αυτοί είναι εστί παρουσία τους. Όμως θα πρέπει να υπάρξει συνένωση δυνάμεων, να βρεθεί μια λύση. Δεν θα φύγει από μόνο του το πρόβλημα αυτομάτως, αν δεν κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ιουμπάμ, Μολδαβία, Ουκρανία. Πολύ επιτυχημένη αποστολή. η διαχείριση των συνόρων νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμη σημαντικότερο καθήκον και όχι μόνο σε αυτά τα σύνορα και γύρω-γύρω. Υπάρχει βέβαια το ζήτημα του Ντομπάς, που είναι ρευστό το καθεστώς του προς το παρόν. Αλλά σε αυτή την περιοχή είτε θα πρέπει η συμβουλευτική αποστολή να ε, επιμηκυνθεί ως προς τη θητεία της, προ την εντολή της. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί ε, η κατάσταση το Σύνταγμα μέχρι τα τέλη του έτους, όπως και τα σύνορα. που είναι κάπως ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να στείλουμε ακόμη κόσμο να ελέγχει τα σύνορα. Οι Ουκρανικές αρχές πρέπει όμως να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τα σύνορα. Άρα χρειάζεται κατάρτιση εξοπλισμό, υποστήριξη κτλ. Πολλά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτός ένας τομέας, είναι μια περιοχή και στρέφομαι και στην ΟΕΜ στο Κίεβο. Απ' την άλλη, άλλη επιλογή είναι η αποχώρηση, η μετακίνηση από την περιοχή, γιατί προς το παρόν περιζόμαστε στο στρατηγικό επίπεδο, παραμένοντας στο Κίεβο δηλαδή. Είναι σημαντικό βέβαια αυτό για να υπάρχει τάξη από εκεί ξεκινάει κανείς, ε, ξεκινάει από το Κίεβο, από πάνω προς τα κάτω. Όμως, οι συνάδελφοί μας, οι Ουκρανοί, ζητούν περισσότερη προβολή επιτόπου, γιατί τώρα πρέπει να κερδίσουν το μυαλό και την καρδιά του μέσου Ουκρανού πολίτη. Άρα τι κάνουμε στην Ουκρανία. Στηρίζουμε τον ΟΑΣΕ που είναι ο βασικός ε, διεθνής παράγοντας ε, που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ αλλά έχουμε και μια αυτόνομη δράση που θα μπορούσε να ε, επεκταθεί και να καλύψει για παράδειγμα τα σύνορα ή την εκπαίδευση της αστυνομίας. στρατηγική εξόδου, στρατηγική μετάβαση κτλ. Ουσιαστικά στόχο έχει να προσπαθήσει να περάσει ένα μήνυμα. Αν έχουμε στην εργαλειοθήκη μας διάφορα μέσα, μεταξύ αυτών ε, ΚΑΠΑ, αλλά και άλλα. Στρατηγικά, μη στρατηγικά, αλλά και ανάπτυξη και άλλα. Η ισχύ της Ένωσης που την καθιστά μοναδική είναι ότι μπορεί να μετακινείται μεταξύ αυτών των εργαλείων, γιατί τα έχει στην εργαλειοθήκη της όλα αυτά. Αυτό δεν ε, το έχει κάποιος άλλος. Μπορεί να πηγαίνω έρχεται κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να αναπτύσσεται αρχικά μια στρατιωτική επιχείρηση, έπειτα αναλαμβάνει πολιτοφυλακή, μια μη, ε, στρατιωτική αποστολή και επανέρχεται μετά στρατιωτική αποστολή για κάποιο λόγο, αν χρειαστεί κτλ. Άρα υπάρχει εναλλαγή στη χρήση των εργαλείων και όταν είναι δυνατόν να δοθούν οι ευθύνε ε, στι τοπική, στις τοπικές αρχές, και αυτός είναι σημαντικός ο στόχος, δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα εξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες να σταθούν στα πόδια τους και να έχουν τη δυνατότητα να κυβερνούν τη χώρα τους με τον σωστό τρόπο. Αυτή είναι η στρατηγική μετάβαση. Κύριε Διευθυντάλη Πρόεδρο, σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να απαντήσετε ίσως τα ερωτήματα του κυρίου Φρόιντ, σύντομα, σύντομα. Και τα δικά μου αφήστε τα, δεν πειράζει, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και κλεισμένα των θυρών με την νομική υπηρεσία. Ο διευθυντής κύριος ε, Ναι, συγγνώμη, για τη Λιβύη και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη πρόσφατη εμπειρία στη Λιβύη, η Ιουμπάμ Λιβύη. Αποσύρθηκε σε εμβριακή κατάσταση διατηρείται ε, εν ζωή. Ε, ουσιαστικά μιλάμε όμως για τρία-τέσσερα άτομα ε, που είναι στην την στην. Αλλά η πρώτη εμπειρία ήταν η εξή. Η απλή και μόνη παροχή εκπαίδευση δεν βοηθάει. Χρειάζεται υλικό εξοπλισμός και πρέπει να ενδιαφερθεί εκεί ο κόσμος πρέπει να πλασάρουμε τα δικά μας συμφέροντα και ίσως να μην φαίνεται και να μην ακούγεται και πολιτικός ορθό αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Το να πας και να τους πεις ότι ήρθαμε να σας διδάξουμε το πώς θα φτιάξετε τη χώρα σας, τι θα κάνετε, πώς θα κάνετε το ένα το άλλο, δεν αρκεί, έχει αποδειχθεί. Πρέπει να προσελκύσουμε, να κινήσουμε το ενδιαφέρον τους. Γι' αυτό στη δημιουργία υποδομών πρέπει να περιλαμβάνεται και εκπαίδευση, αλλά και η παροχή υλικού εξοπλισμού. Αυτά ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Δευθύντα. Πολύ μεγάλη συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό. Παρακαλώ τους συναδέλφους να μην αποχωρήσουν. Έχουμε και κλεισμένο των θερών των θυρών συνεδρίαση μόνο για βουλευτές, πολιτικούς συμβούλους, πολιτικών ομάδων, γραμματεία. Οι λοιποί παρακαλώ να αποχωρήσουν. Thank you, Director. Thank you, Madam Chair. Thank, you. very much. At any time, really. <laughs> Please leave your headphones. Oh, oh, oh, yeah. <laughs> It may